Welcome back for the afternoon session. Καλώς επιστρέψατε στην απογευματινή συνεδρίαση και να ξεκινήσω με τα συμπεράσματα της συνάντησης των συντονιστών που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί. Υιοθετήσαμε την τροποποιημένο σχέδιο ημερήσιας διάταξη τη συνάντησης τη 10 και 11 Οκτωβρίου. Για το σημείο 2 δεν έχουμε να αναφέρουμε γνωμοδοτήσεις ή εκθέσεις για τις αμφισβητούμενες συστάσεις που ε, απασχόλησαν μεγάλο κομμάτι της συνάντησης. Υιοθέτησα εγώ, ε, υιοθέτηθηκαν οι συμβιβασμοί μου για τρεις ε, αναφορές 0211, 0213 και 0243 και για την 0249 του 2016 η συμβιβαστική μου εγκρίθηκε με μια προσθήκη να τη στείλουμε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς ενημέρωση για το αίτημα που αφορούσε τα σημεία Β που υπήρχαν αρχικά στην λίστα Β του Ιουνίου. Ορισμένα έκλεισαν και ξέρω ότι θα βαρεθείτε αυτά που σας λέω αλλά πρέπει να τα διαβάσω για να περαστούν στα πρακτικά. του 11, 0357 του 12 και 2214 του 14 η απόφαση για να κλειστεί αυτή η αναφορά έγινε με ψηφοφορία μετά από ανταλλαγή απόψεων. Το αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας ήταν 20 υπέρ του κλεισίματος της αναφοράς και 14 υπέρ του να διατηρηθεί ανοιχτή. Στη συνέχεια, ε, επειδή έφτασαν νέες πληροφορίες, οι ακόλουθες αναφορές παραμένουν ανοιχτές για περαιτέρω διαρεύνηση επειδή λάβαμε πληροφορίες μόλις χθες. Πρόκειται για, τις, για την 0355 του 10 και για την 1342 του 11. Τα σημεία της λίστας Β του Ιουλίου για τα οποία είχε προταθεί προς την παρακολούθηση τα εξή μάλλον θα παραμένουν ανοιχτά και θα ε, αναλυφθεί η συγκεκριμένη δράση όσον αφορά τις αναφορές τις αναφορές 0254 067 099, 0461, 08, 07. Η 0467 θα κλείσει αφού εστάλει η επιστολή στην άκρη και αφού αυτό γίνει έχουμε συμφωνήσει να κλείσει τρεις αναφορές η 0165 η 2299 και η 0549 έκλεισαν για το σημείο 5 που αφορά το χρονοδιάγραμμα συναντήσεων του 2017 της Επιτροπής αυτής. Το ημερολόγιο εγκρίθηκε. Στο σημείο 6 η αρχή που αφορά τη συμμετοχή τρίτων ατόμων πέραν των ε, όσων έχουν υποβάλει αναφορές και εκείνων που εκπροσωπούν ε, τις δημόσιες αρχές τις οποίες αφορούν αναφορές ε, ανταλλάξαμε απόψεις και συμφωνήσαμε να τηρηθούν απόλυτα οι καθηθυντήριες οδηγίες επί του θέματος δηλαδή με άλλα λόγια πριν καλέσουμε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο θα πρέπει να προηγηθεί η συμφωνία των συντονιστών. Για το σημείο 7, σχεδιασμός του πρώτου κομματιού του 2017, που αφορά τις δημόσιες ακροάσεις και τις επισκέψεις αντιπροσωπιών, κλήθηκαν οι ομάδες να συντονίσουν τις προτάσεις τους μεταξύ τους, μεταξύ των ομάδων, για διερευνητικές επισκέψεις και ακροάσεις στο πρώτο εξάμεινο του 2017, ώστε τον Οκτώβριο, στις 11 Οκτωβρίου η απόφαση ε, να μπορεί να ληφθεί και ε, το πολύ δύο επισκέψεις και δύο ακροάσεις για το σημείο 8 η επερχόμενη διερευνητική αποστολή επίσκεψη στη Σλοβακία που θα λάβει τώρα 22-23 ε, Σεπτεμβρίου χώρα και στο Τάραντο στην Ιταλία από τις 2 μέχρι τις 4 Νοεμβρίου οι συντονιστές ενέκριναν το πρόγραμμα και το κατάλογο συμμετοχόντων ε, ε, στη Σλοβακία και το προκαταρκτικό πρόγραμμα για την επισκέψη στο Τάραντο στην Ιταλία. Στο σημείο 9 το ενημερωμένο σχέδιο προγράμματος για την οκρόαση που αφορά τα εμπόδια στην ε, μετακίνηση, στην κυκλοφορία και στην εργασία των πολιτών στην ευρωπαϊκή αγορά όπως, υποβλήθηκε από τους αναφορά. Οι συντονιστές Ενέκρινα το πρόγραμμα για την ακρόαση και μετά την παρακολούθηση της ηλιακής ενέργειας ε, όσον αφορά τις ε, συζητήσεις περί αναφορών και έχουμε πολλές τέτοιες αποφασίσαμε να προβούμε σε ένα ε, σύντομο ψήφισμα επί του θέματος. Θα συνταχθεί ένα σχέδιο για τη συνάντηση του Νοεμβρίου με σκοπό να υιοθετηθεί το κείμενο στην Επιτροπή τον Ιανουαρίου του 2017. Σημείο 11 αφορά τις αναφορές για το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου και τα σχετικά ζητήματα. Εγώ ενημέρωσα τους συντονιστές για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις αναφορές για το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 10 η ενδιάμεση αναθεώρηση του ετήσιου ε, προγράμματος έρευνας του Τμήματος Πολιτικής ΣΥ. Οι συντονιστές ε, ε, έλαβαν γνώση του εγγράφου. Το σημείο 13 αφορούσε την αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού και οι συντονιστές συμφώνησαν να υποβάλουν από κοινού ε, τροπολογίε στην έκθεση Κόρμπιτ ε, για τον εσωτερικό κανονισμό. Και συμφώνησαν άπαντες για την αποφάση αυτή. Ε, τώρα τα σημεία ενημέρωσης Έλαβα γνώση οι συντονιστέ και έτσι κλείνει, έκλεισε η συνεδρία των συντονιστών. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαριά για μια πολύ σύντομη δήλωση. How brief is brief. Πόσο σύντομο είναι σύντομο. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, όπως είπα και κατά την ε, συζήτηση των συντονιστών, η απόφαση η οποία ελήφθη να απορρίψει την ένσταση που είχα υποβάλει στις 27 Πέμπτου προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ΠΑΕΑ ΔΟΣΟΕ για τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι και νομικά αστήριχτη και πολιτικά απαράδεκτη. Διότι η αναφορά αυτή, όπως θυμόσαστε, τον ε, περασμένο Οκτώβρη, παρότι υπήρχε αντίθετη εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από εισήγηση δική μου έγινε δεκτό από τους συντονιστές να κριθεί ως παραδεκτή. Και απεστάλησαν επιστολές στην Κομισιόν, στην ελληνική κυβέρνηση και στην ε, ε, γερμανική κυβέρνηση. Και εν συνεχεία υπήρξε η άποψη της Κομισιόν η οποία θεωρεί ότι δήθεν το θέμα είναι διμερές και δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούσε επί του πρακτέου ε, να μην υπάρχει καμία τοποθέτηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω ένιπτε τα σχέδια τη σαν πόντιο πιλάτο. Εξηγήσαμε πολλέ φορέ ότι υπάρχει άμεση σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την υπόθεση αυτή. Πρώτον, διότι δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από την απόφαση τη ε, διάσκεψη ειρήνη του 1946 των Παρισίων για τι πολεμικέ επανορθώσει. Δεύτερον, έχει άμεση σχέση διότι καταβολή και εξόφληση των πολεμικών επανορθώσεων και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου είναι βέβαιο ότι αλλάζει τη δημοσιονομική θέση της χώρας επομένως έχει άμεση σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς η ελλάδα θα τεθεί εκτός ε, επιτήρησης. Επιπλέον η Ελλάδα και η Γερμανία δεν έχουν συνάψει καν συμφωνία ειρήνης μεταξύ τους και αυτό είναι θέμα που αφορά δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι έπρεπε η υπόθεση αυτή να μείνει ανοιχτή και ευχαριστώ τους συναδέλφους οι οποίοι ψήφισαν την πρότασή μου, 14 ψήφους πήρε, αλλά βεβαίω η απόφαση να ληφθεί που ελήφθη να κλείσει η υπόθεση είναι υπόθεση η οποία έχει ήδη δημιουργήσει αγανάκτηση στον ελληνικό λαό. Σα μεταφέρω τα συναισθήματα που υπάρχουν από το πρωί που έγινε δεκτή και τεράστια φυσικά απαγοήτευση από αυτού που αισθανόταν ότι κάτι μπορούσε να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όπως σας ενημέρωσα θα υποβάλω νέα αναφορά, θα υποβάλω εγώ ο ίδιος αυτή τη φορά. Δεύτερον, θα ζητήσω να πάει με τη διαδικασία κατεπήγοντος και τρίτον, θα τεθεί ξανά το θέμα αυτό μαζί και με άλλα επιχειρήματα. Και αν απορριφθεί, θα προσφύγω και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τέλος, να επισημάνω ότι η απόφαση αυτή που έλαβαν η πλειοψηφία των συντονιστών, δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους φυσικά βρήκανε στήριγμα ή μάλλον θα έλεγα ότι βρήκαν ευκαιρία από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Διότι ειδοποιήσαμε την ελληνική κυβέρνηση έντονα και έγκαιρα να έρθει να παραστεί σε αυτή την υπόθεση. Να στείλει φάκελο, να υποστηρίξει την υπόθεση των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ενώ ενημερώθηκε η Ελληνική Βουλή στις 27 έκτου Επίσημα δεν το έπραξε. Την προηγούμενη Πέμπτη ενημέρωσα τον κύριο Βούτσι. Και έρχεται η Ελλάδα, δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση, χτες 6 παρα 10 το βράδυ να στείλει τι, το πόρισμα της Επιτροπής της Διακομματικής στα ελληνικά, ένα κείμενο δύο παραγράφων, πότε όταν είχε λήξει η προθεσμία, διότι ξέρουμε ότι τη Δευτέρα έληξε η προθεσμία και εγώ υπέβαλα νέα στοιχεία την προηγούμενη Δευτέρα, και φυσικά με αυτή τη συμπεριφορά κατέδειξε ότι δεν ήθελε να στηρίξει εν προκειμένου αυτή την υπόθεση. Και έτσι πήραν θάρρος διάφορες πολιτικές δυνάμεις να απορρίψουν την έσταση. Και τι ζητούσαμε κυρία Πρόεδρε και τελειώνω. Ζητούσαμε με την έστασή μας πρώτον να μείνει ανοιχτή υπόθεση, δεύτερον να σταλεί επιστολή στην Ελλάδα και στη Γερμανία να έρθουν να τοποθετηθούν επί των ετοιμάτων των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και τρίτον να τοποθετηθεί η Κομισιόν για το τι σχέση και δεσμεύσεις έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη συνθήκη ειρήνης του 1946. Και σας είπα, εν προκειμένου, ότι πώς γνωρίζετε την απάντηση της Γερμανίας. Πώς κλείνετε την υπόθεση πριν έρθουν οι απαντήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν δεκτές. Ο επομένως, κυρία Πρόεδρε, αυτά θέλω να καταγραφούν στα πρακτικά και επισημαίνω για άλλη μια φορά ότι είναι απαράδεκτη η απόφαση η οποία έχει ληφθεί και με την οποία βεβαίως διαφωνώ. Ευχαριστώ πολύ. You Όπως γνωρίζετε δεν ήθελα να ξαναρχίσει αυτή η συζήτηση διότι ελήφθη απόφαση από τους συντονιστές ε, να κλείσει αυτό το ζήτημα και μάλιστα διεξήχθη η ψηφοφορία όπως ε, προβλέπουν ε, οι εσωτερικοί μας κανονισμοί. Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο να ξαναρχίσουμε να συζητούμε το θέμα στην παρούσα χρονική στιγμή. Κυρία Σακοράφα, κυρία Κούνεβα, σα ερωτώ πραγματικά, είναι απαραίτητο, θεωρείτε τώρα να το ξανασυζητήσουμε από τη στιγμή που με την ψήφο του, οι συντονιστέ αποφάσισαν να κλείσει αυτή η αναφορά. Κύριε Σακοράφα, αλλά προσπαθήστε να είστε σύντομοι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό για όλου εμά του Έλληνε. Εγώ μία δήλωση θέλω να κάνω, του ενό λεπτού δεν θα σα καθυστερήσω ούτε θα ταλαιπωρήσω την Ε, ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Θέλω να απευθυνθώ προς εσάς, προς το Προεδρείο και τους αγαπητούς συναδέλφους. Κυρίες συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι σήμερα σε αυτή την αίθουσα θα δόθηκαν νομικές τεκμηριώσεις, διασταλτικές ερμηνείας περί αρμοδιοτήτων για ένα ζήτημα όμως που θέλω να το περιγράψω με την ακρίβεια του βάρους που έχει. Μιλάμε για τις αξιώσεις που συνδέονται με τα πιο ιδεχθή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και προκειμένου κατά του ελληνικού λαού. Αξιώσει απαράγραπτε από την ιστορία, την πολιτική αλλά και την αδυναμία, τη δικονομία. Περί αυτού πρόκειται η όποια προσπάθεια υποβάθμισή του σε ερμηνείε υποκρύπτει την πλήρη συνθηκολόγηση τη Ευρώπη των αξιών στο κυρίαρχο ευρωπαϊκό κατεστημένο που παραμορφώνει την ιστορία και αγνοεί επιδεικτικά τι πληγέ που προκάλεσε στο λαό μα μια άλλη ιστορική στιγμή αυτή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιστορία όμω που δεν δικαιώνεται ποτέ δεν κλείνει και με την έννοια αυτή το ελάχιστο που θα έπρεπε να έχει γίνει είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά όπως επιτάσσει το δίκαιο, η δικαιοσύνη, η ηθική και η πολιτική υποχρέωση που έχει η σύγχρονη Ευρώπη και η σύγχρονη ευρωπαϊκή λαή σε αυτούς που αντιστάθηκαν στον ναζισμό. Αυτό δεν αποτελεί χρέο μόνο στην ιστορία, αλλά και χρέο απέναντι στο ποτέ ξανά. Αυτά κυρία Πρόεδρε και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κούνεβα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ε, επίσης και εγώ θέλω να μην κλείσει αυτό το θέμα. Πρέπει να μένει ανοιχτό και να το συζητήσουμε σοβαρά. Εμείς οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η ευρωομάδα της ΓΟΕ πιστεύουμε ότι το θέμα των πολεμικών οφείλων της Ελλάδας δεν πρέπει να τεθεί στο αρχείο πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή μας. Με αφορμή τις αναφορές που κατατίθενται στην Επιτροπή Αναφορών από πολίτε και φορείς οι οποίοι ζητούν να εξεταστεί το θέμα των γερμανικών οφειλών προ την Ελλάδα παίρνουν το λόγο για να ενημερώσουν τα μέλη τη Επιτροπή Αναφορών ότι ο πρόεδρο τη Ελληνικής Βουλή ενημέρωσε με επιστολή την πρόεδρο τη Επιτροπή και το και τους συντονιστές για τις θέσεις της ελληνικής Βουλής και της ελληνικής κυβερνήσης αναφορικά με αυτό το μέγα θέμα. Θέμα μεγάλη πολιτική, ιστορική και δικαιακή σημασία, το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή Αναφορών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής απέστειλε επίσης το πόρισμα της ε, Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για την διεκδίκηση των γερμανικών κατοχών οφειλών, το πόρισμα θα συζητηθεί σύντομα στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική και σχέδια για το θέμα. Όπως είπε και πρόσφατα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπαρας, επιτιμούμε να κλείσουμε επιτέλους αυτή την ανοιχτή πληγή στο σώμα της δικαιοσύνης, στο ίδιο το σώμα της, Ευρώπη. της Ευρώπης. ευχαριστώ. Okay. Um, Μάλιστα. Να κάνω κάποιες διευκρινήσεις σε αυτή τη φάση. Και σας παρακαλώ να προσέξετε το εξής. Στο παρόν στάδιο δεν είναι το θέμα καθόλου η παραδεκτότητα, το αν είναι παραδεκτή ή όχι η οχι αυτή. Πρόκειται για μια απόφαση που αφορά είτε να κλείσετε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μετά από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή την απόφαση κλήθηκαμε να λάβουμε. Υπάρχει ένα non-paper, έναν επίσημο έγγραφο που υπευλήθη στην Επιτροπή μας τον Ιανουάριο του 2015 από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, στο οποίο διαβάζω λέει ότι οι πολεμικές επανορθώσεις ε, από τις ε, ζημιές ε, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου δεν μπορεί ε, ως θέμα να συνδεθεί με καμία από τις συνθήκες Ευρωπαϊκής, από τις διατάξεις των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει των άρθρων 2 έω 6 των συνθήκων. Ούτε μπορεί το θέμα αυτό να θεωρηθεί ότι είναι στόχος της Ένωσης, όπως αυτοί που περιγράφονται στο άρθρο 3 των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ουδέποτε ανεμίχθη σε οδήποτε δραστηριότητα σχετική με επανορθώσεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπλέον, το συμπέρασμα πρέπει να είναι ότι η Ελλάδα τα θέματα, οι σχέσεις και οι αξιώσεις, οι διεκδικήσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας αφορούν αποκλειστικά τις διμερείς σχέσεις των δύο λόγω κρατών. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν συμφώνως προς τις ισχύουσες διατάξεις ε, του διεθνούς δικαίου. Κατά συνέπεια, το όλο αυτό ζήτημα είναι εκτός πεδίου αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εκτός δικαίου, δεν εμπίπτει στο ε, πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ ε, λίγη παραπομπή μου στην απάντηση της νομικής υπηρεσίας. Βέβαια, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου το θέμα. Να γίνει μια δίκη. Μπορεί κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο για αυτό το θέμα. Και θα το έλεγα σε κάθε αναφέροντα το ίδιο. Εάν θεωρείτε, αναφέροντας ότι έχετε το δικαίωμα, θεωρείτε ότι η αναφορά σας δεν αντιμετωπίστηκε με το δέοντα τρόπο, παρακαλώ πηγαίνετε στο δικαστήριο. Και το ίδιο έχω να πω και για την προκειμένη αυτή υπόθεση. Πέραν των τύπων, εγώ πρέπει να πω ότι προσωπικά, και νομίζω όλοι μας εδώ στην αίθουσα, πραγματικά νιώθουμε ε, μεγάλη συμπαράσταση και συμπάσχουμε με τον ελληνικό λαό. Εμένα ραγίζει η καρδιά μου ε, να βλέπω ότι εξακολουθούν να υποφέρουν οι Έλληνες πολίτες ακόμη και σήμερα. Όμως, όμως πρέπει να εμείνουμε στις αρχές και στις αρμοδιότητες και εδώ μιλώ νομίζω ε, ως εκπρόσωπος του παρόντος θεσμικού οργάνου που ούτε αυτό ούτε κανένα άλλο θεσμικό όργανο δεν ασχολήθηκε με μια ανάλογη υπόθεση κατά το παρελθόν. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να βάζουμε ένα νέο πολιτικό αποτύπωμα, ένα νέο ίχνος να αφήνουμε και δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πρέπει να τηρήσουμε τις συνθήκες που έχουμε ως πλαίσιο. Ελπίζω κύριε Μαριά να καταλαβαίνετε ότι κανένας ε, δεν θέλει το κακό των Ελλήνων. Όλοι θέλουμε το καλό της χώρας, την ευημερία της χώρας, αλλά με αυτό και αυτό θέλω να κλείσω τη συζήτηση ε, για την αναφορά που θεωρώ ότι πρέπει να κλείσει και περνάμε στο σημείο 11 της μερίσιας διάταξης που είναι η τίσια έκθεση για τις δραστηριότητες ε, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2015. Νομίζω ότι είναι σημαντικό θέμα αυτό, πρέπει να το συζητήσουμε με το δέοντα τρόπο, η συγκεκριτή ε, ορίστηκε στη συνεδρίαση των συντονιστών ε, του Μαρτίου του 2016 ο κύριος Μαριά, ο οποίος θα μα παρουσιάσει την έκθεσή του. I'm Σας δίνω το λόγο με τα χαρά για αυτό το θέμα, κύριε Μαριά. Έχω κυρία Πρόεδρε. Για να υπολογίσω την ομιλία. Περίπου, περίπου πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, θα παρουσιάσω την ε, ε, εισήγησή μου για το θέμα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αυτό που έχει σημασία είναι βεβαίως να δούμε το πώς μπορεί να δουλέψει ένα όργανο όπως είναι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και να αντιληφθούμε ότι τα μη δικαιοδοτικά όργανα όπως είναι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αλλά και η Επιτροπή Αναφορών έχουν τη δυνατότητα να διερευνούν υποθέσεις βεβαίως πάντοτε εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων τους αλλά με τρόπο ο οποίος να μην είναι πολιτικά φορτισμένος. Διότι επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε, όπως ανακοινώσατε προηγουμένως την απόφαση και τη διαβάσατε, οι τελευταίες σας λέξεις απέδειξαν ότι ήταν πολιτικά φορτισμένη η απόφαση της Επιτροπής Αναφορών των συντονιστών της για τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις. Γιατί είπατε δεν μπορεί να κάνει αυτό το βήμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ σας λέω θα το κάνει κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν τα, δικαιο... τα μη δικαιοδοτικά όργανα σε διαφορά με τα δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν παραπέρα, να ανοίξουν δρόμους. Και χαίρομαι που στην περίπτωση του Όμπουτσμαν ή της Όμπουτσγούμαν για την ακρίβεια, της κυρίας Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο κινείται εντός των πλαισίων του κανονισμού, αλλά έχει ευρύ πνεύμα, βλέπει μακριά, δεν έχει φόβο και ανοίγει δρόμους. Παράδειγμα, θεωρώ πολύ σημαντική την τοποθέτηση που έκανε για την περίπτωση του κυρίου Μπαρόζο Δηλαδή αυτό που ονομάζει revolving doors. Δηλαδή το να είναι κάποιος επίτροπος και εν συνεχεία να παίρνει ένα πόστο σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Και αυτό που έκανε με μεγάλο θάρρος αυτές τις μέρες και κατέδειξε ότι δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος της Κομισιόν και ταυτόχρονα να γίνεσαι πρόεδρος αργότερα ενός, να, να εργάζεσαι μάλλον σε ένα πολύ συγκεκριμένο οργανισμό όπως ήταν η Goldman Sachs. Άρα λοιπόν τι θέλω να πω ότι στην έκθεσή μου και βεβαίως την έχετε μπροστά σας και θα ακούσω ε, με χαρά τους συναδέλφους να κάνουν τις παρατηρήσεις τους ούτω ώστε να δημιουργήσουν μια συνθετική άποψη για να μπορέσουμε να έχουμε μια έκθεση καλή, να γίνουν αποδεκτές βεβαίως και οι τροπολογίες. Αλλά το βασικό είναι ότι αυτό το όργανο αποδεικνύει ότι ως διαμεσολαβητής μπορεί και βλέπει μακριά και μπορεί να προλαβαίνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία αυτή τη έκθεση. Πρώτο, ένα θέμα διαφάνεια. Τι θα γίνει με την λειτουργία τη ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της Κομισιόν, αλλά και των άλλων οργάνων. Υπάρχει διαφάνεια στην, περίπτωση στην περίφημη TTIP. Πώ γίνονται εκεί οι διαπραγματεύσει, Αυτά λοιπόν τα έθιξε η έκθεση και νομίζω ότι τα έβαλε με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Διότι εκεί Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Επόμενο θέμα. Τι γίνεται με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Μήπως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μόνο νομισματική αρχή. Είναι όμως και μέλος της Τρόικας. Είναι και δανειστής κάποιων κρατών. Μήπως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στη λειτουργία της. Αυτό το θέμα επίσης θίγεται και έχει ενδιαφέρον. Τι γίνεται με το ρόλο των, της ίδιας της Κομισιόν. Μήπως και αυτή στο πλαίσιο του Μνημονίου και της Τρόικας έχει σύγκρουση συμφερόντων. Άρα λοιπόν αυτά τα μεγάλα ζητήματα νομίζω ότι τίθενται, όπως βεβαίω τίθενται ζητήματα που είχαν θέσει προηγούμενες εκθέσεις, στις οποίες αναφέρθηκα, όπως η έκθεση που είχε κάνει ο κύριος Βαλέσα την πρώτη χρονιά και η επόμενη χρονιά που ήταν από τη συνάδελφο της ε, σοσιαλιστικής ομάδας. Δηλαδή κρατούμε τα συμπεράσματα των εκθέσεων που έκαναν οι συνάδελφοι και προσπαθούμε πάνω στα συμπεράσματα αυτά σε συνδυασμό με τις νέες προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν να κάνουμε προτάσεις. Επίσης, τι γίνεται με την περίφημη πρωτοβουλία των πολιτών, όπου πρέπει να αναπτυχθούν τα ζητήματα. Υπήρχε πρωτοβουλία για τα θέματα του νερού, η οποία θαύτηκε με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν κυρία Πρόεδρε νομίζω ότι τα βασικά σημεία της έκθεσης υπάρχουν. Περιμένω τους συναδέλφους να κάνουν παρατηρήσεις. Δεν θα εξαντλήσω τα πέντε λεπτά. Θα μείνω εδώ. Αναμένω τις παρατηρήσεις και μετά όταν τελειώσουν οι συνάδελφοι, αν έχω ένα λεπτό, να πω μια ε, κεντρική κουβέντα για να συμπεράνουμε το πού μπορούμε να καταλήξουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ εγώ εσάς, κύριε Μαριά. Δεν ζητάει κανείς το λόγο. Α, κυρία Πιτέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια επικεντρώθηκε κυρίως στην διαφάνεια και διάφορα θέματα που συνδέονται με αυτήν. Έχω διάφορες παρατηρήσεις που ίσως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο κείμενο. Μιλώ ως ε, κάποιο που έχει πείρα και από τις δύο πλευρές, διότι για ένα διάστημα ήμουνα μέλος της πολωνικής ομάδας για τη διαφάνεια. Όσον αφορά τα δημόσια έγγραφα, μόλις είχαμε εισάγει στην Πολωνία νέα, νέο νόμο για το θέμα αυτό και Εργάστηκα και στην κυβέρνηση του Ντόναλτ Τούσκ όταν ήταν ε, Πρωθυπουργό. Έχω λοιπόν πείρα και από την κυβέρνηση. Μπορώ να πω το εξής όλα τα θέματα που συνδέονται με τη διαφάνεια έχουν και κάποια όρια. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για να στηρίξω αυτό το επιχείρημα, ιδιαίτερα στον δημόσιο χώρο. Για παράδειγμα, οι διαπραγματευτές για διεθνείς συμφωνίες. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημοσιεύει την διαπραγματευτική του θέση πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων, διότι αυτό θα αποδυναμώσει την διαπραγματευτική του θέση. Δεύτερον, όπου υπάρχουν συγκρούσεις σε υποθέσεις στα δικαστήρια. Είναι πάλι δύσκολο φανταστούμε να δημοσιευτούν όλες οι θέσει ε, πριν την έναρξη της δικαστικής διαδικασία Και υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα. Ξέρω ότι ο εισηγητή ε, θέλει να επικεντρωθεί στην ε, διαφάνεια και την κοινοποίηση, την αποκάλυψη δημοσίων εγγράφων, αλλά ποια είναι τα όρια που θα θέσουμε, διότι κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να ισχύει η διαφάνεια χωρίς όρια. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο σαν σύνθημα, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε και τα πολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι ακόμα. Έχουμε την ε, περίπτωση αποζημίωσης επανορθώσεων. Ε, ένα κράτος μέλος ε, θα θέλει να αποκαλύψει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Και αυτό που λέτε για τις περιστρεφόμενες πόρτες, ε, πιστεύετε ότι όλα έχουν γίνει θελημένα. Νομίζω ότι πρέπει να δηλώνουμε τα ονόματα που γνωρίζουμε, αλλά στην περίπτωση αυτή φαίνεται μάλλον σαν να θέλουμε να κατηγορήσουμε ένα άτομο αντί να λύσουμε το πρόβλημα των ε, περιστρεφόμενων ε, θυρών. Θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε το θέμα ή απλά θέλουμε να βρούμε κάποιον να κατηγορήσουμε. Πιστεύω ότι το έγγραφό μας ε, θα πρέπει να δείξει τον τρόπο να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Τζουντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δυστυχώ η σκιώδη εισηγήτρια Μιριαμ Ντάλι δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα, αλλά μου ζήτησε να ε, διαβάσω μια σύντομη δήλωση. Η Μίριαμ θέλει να συγχαρεί τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του που τονίζει τα πιο σημαντικά ε, μέρη της εργασίας της διαμεσολαβήτριας και προσβλέπει στις διαπραγματεύσεις με τον εισηγητή. Η Μίριαμ θέλει να τονιστούν ακόμα περισσότερο οι εργασίε τη διαμεσολαβήτρια, ιδιαίτερα στον χώρο των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στην περίπτωση των Ταμείων Συνοχής. Η έρευνά τη έδειξε διάφορες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν Ταμεία Συνοχής για να χρηματοδοτηθεί η διατήρηση σε ιδρύματα παιδιών αντί να γίνει μετάβαση σε υπηρεσίες που προσφέρονται από την κοινότητα. Αυτές οι μικρές προσπάθειες ε, κάνουν μεγάλη διαφορά στις ε, καθημερινές ζωές των πολιτών. Είναι λοιπόν σημαντικό να τονίσουμε τις προσπάθειές της ε, σε αυτόν τον τομέα. Η σκιώδη εισηγήτρια πιστεύει επίση ότι η δουλειά τη διαμεσολαβήτρια ε, στο να προστατεύει ε, του whistleblowers είναι πολύ σημαντική. Η Μίρια με τονίζει ότι με έρευνά της η διαμεσολαβήτρια ε, βρήκε ότι 7 από 9 θεσμούς δεν συμμορφώνονται με ε, τους σχετικούς κανόνες. Ε, ένα από τα 7 θεσμικά όργανα ε, που δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η σκιώδη συζήτρια πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να τονιστεί στην έκθεση που να δείχνει ακριβώς ότι είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ο κ. Τερικαπράς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, η έκθεση είναι εξαιρετική. Πρέπει να τον αναγνωρίσουμε και να συγχαρούμε την κυρία Εμιλιορέλη. Εξαιρετική αναφορά. Δεδομένου αυτού, δύο σχόλια τώρα για τη διαφάνεια. Λυπούμαστε ιδιαίτερα το ότι όλο και περισσότερο γίνεται πραγματικότητα οι αίθουσε ανάγνωση, όπως για το TTIP ε, και για τα γενετικώς τροποποιημένα για τα μεταλλαγμένα, για τα GMO. Ε, δεν λειτουργεί όλο αυτό υπέρ της διαφάνειας, το να κρύβουμε από τους ευρωβουλευτές, ακόμη και από τους ευρωβουλευτές τα όσα συμβαίνουν. Τρίτον, τρίτο σημείο, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να ενημερώνουμε τους πολίτες για το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Το θέμα είναι να ερμηνεύσουμε το αρθρό 51 με λιγότερο περιοριστικό τρόπο. Στην ΠΕΤΗ είχε λάβει η χώρα τον περασμένο Μάρτιο μία ακρόαση για το θέμα αυτό. Και ο απότερος σκοπός ε, αυτής της νέας ερμηνείας θα πρέπει να είναι να, η, απαλήψη, η αυτού του αρθρού 51 κατά την απόψή μου. Τώρα όσον αφορά τις περιστραφόμενες πόρτες νομίζω ότι πρέπει να μεριμνήσουμε για την πρόληψη και την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων. Δεν μπορεί να μας αφήνει ίσχους μια κατάσταση κάποιος ο οποίος κάνει ένα λάθος και μετά λέει λυπάμαι και το μετανιώνω. η ακολουθία αμάρτημα ε, και συγγνώμη πρέπει να αποφεύγεται ε, όσο το δυνατόν περισσότερο στη δική μας ε, ηθική συμπεριφορά γιατί δεν αρκεί δεν υπήρχε λάθος και δεν υπήρχε αμάρτημα δεν υπήρχε λόγος και για να ζητήσει κανείς συγγνώμη θέλουμε να αναθεωρηθεί ο κώδικας διοντολογίας της Κομισιόν και όλοι οι κώδικες διοντολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γι' αυτό το σκοπό πιστεύω ότι πρέπει να καταστήσουμε υποχρεωτικό τον κώδικα ε, χρηστής συμπεριφορά συμπεριφοράς που σχετίζεται στενά με ε, τις δραστηριότητες του Δημοσιολαβητή. Ευχαριστώ κύριε Τερικαμπράς και δίνω το λόγο στην Ελεονόρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Νότι Μαριά για το κείμενο αυτό το οποίο κατά την απόψή μου αγγίζει θέματα κλειδιά στα οποία έχει επικεντρωθεί η θεσμική δράση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβητή ε, και πάει και πιο πέρα από αυτά. Είναι σημαντικό λοιπόν όπως είπε πριν από λίγο ο συνάδελφος η νομοθετική και πολιτική δραστηριότητα τέτοιων προσώπων είναι σημαντική. Πολύ σημαντική και κυρίως ε, για αυτό που παίζεται αυτή τη στιγμή ε, σε τέτοιες ιστορικές εποχές η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου δεν συμφωνώ με κάποιες θέσεις. Όσον αφορά τις περιστρεφόμενες πόρτες, για παράδειγμα, είναι ένα σημαντικό μήνυμα το να συμπεριλάβουμε μια από τις πλέον τρανταχτές ε, υποθέσεις τελευταία ε, στη ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υπόθεση ε, Μπαρόζο. Ναι, συμφωνώ να υπάρχει ένα ισχυρό μήνυμα γιατί αυτές οι πρακτικές διαπράττονται ακόμη εντός των θεσμικών οργάνων και σήμερα. Επίσης είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να μιλάμε για έλλειμμα διαφάνειας διότι στην Ευρώπη αυτό ζούμε ένα έλλειμμα διαφάνειας σε πολλούς χώρους όπως βλέπουμε όπω αυτού με του οποίου ασχολείται η Ευρωπαϊκή Δημοσιολαβήτρια ήδη, αλλά και σε άλλου, όπω αναφέρθηκε προηγουμένω, η χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων, για παράδειγμα, εγώ σκέφτομαι, έχω στο και τα μεγάλα έργα τα οποία πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και ειδικότερα εκείνα που είναι διασυνοριακά και τα οποία εξακολουθούν και για τα οποία εξακολουθεί να υπάρχει πολύ περιορισμένη πρόσβαση από τους πολίτες ε, στα σχετικά έγγραφα ε, αλλά και από τους ερετούς ε, και από τους ευρωβουλευτές για παράδειγμα. Οπότε έχουμε ένα έλλειμμα διαφάνειας το οποίο πρέπει να επιληθεί. Επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο σχετίζεται με όλα αυτά είναι η διαρκής και μόνιμη παρουσία των βιομηχανικών συμφερόντων εδώ σε αυτά τα θεσμικά όργανα, δηλαδή η παρουσία των λόμπι εδώ όπου για παράδειγμα ένα υποχρεωτικό μητρό διαφάνειας είναι κάτι που ακόμη δεν συζητείται καν. Δεν έχει συμπεριληφθεί σε καμία ημερήσια διάταξη αυτών των θεσμικών οργάνων. Υπάρχουν πολλά λοιπόν να γίνουν και η δουλειά τη διαμεσολαβήτρια είναι θεμελιώδη σημασία. Και εμεί με αυτέ τι εκθέσει μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε η έκθεση αυτή να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται ο κατάλογος ομιλητών. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 26 Σεπτεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίας. Θέλετε να ξαναπάρετε το λόγο, κύριε Μαριά, παρακαλώ. Ε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις που έκαναν προκειμένου να βελτιώσουμε την έκθεση. Ε, πολλά θέματα τα οποία τέθηκαν πραγματικά θα τα λάβω υπόψη τους ώστε να μπορούμε ε, να καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία να έχει την ε, μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη. Μία μόνο παρατήρηση να πω στη συνάδελφο του, του ΕΛΚ. Ε, όταν ζητούμε διαφάνεια κατά τις διαπραγματεύσεις για την TTIP, αυτές έχουν την έννοια της ενημέρωσης των ίδιων των βουλευτών. Διότι όταν η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, σημαίνει ότι απέναντι πλευρά οι ΗΠΑ γνωρίζουν τις θέσεις Ευρώπης. Εμεί θέλουμε οι βουλευτές να γνωρίζουν επίσης τις θέσεις τις δικέ μας. Οι δικοί μας βουλευτές. Άρα λοιπόν εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολύ δε περισσότερο όταν μας πάνε σε ένα γραφείο που δεν μπορούμε να κρατήσουμε σημειώσεις, που δεν μπορούμε να έχουμε την ευχέρεια να προετοιμαστούμε, διότι εκεί δεν επιτρέπεται να κρατάς σημειώσει στη, στην TTIP. Το ξέρετε αυτό. Όταν πας σε ένα ειδικό γραφείο για να δεις τα έγγραφα της TTIP, φίλε ε, Βαλέσα, δεν επιτρέπεται να κρατάς σημειώσεις, δεν επιτρέπεται να έχεις το κινητό μαζί σου και πρέπει εσύ ως βουλευτής να έχεις την τεράστια δυνατότητα να θυμάσαι τα πάντα. Για ποιο λόγο. Να σε ενημερώσω δε, φίλε συνάδελφε Βαλέσα, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός για τους γερουσιαστές. Οι γερουσιαστές έχουν τη δυνατότητα να δουν όλα τα έγγραφα. Το ίδιο και οι βοηθοί, βοηθοί τους. Και δεν υπάρχει και υποχρέωση χεμήθειας. Άρα λοιπόν δέστε τα αυτά τα θέματα, πάμε να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Εμείς μιλούμε για διαφάνεια σε σχέση με τα έγγραφα που πρέπει να λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα νομοθετήσει και που πρέπει να παρακολουθεί τη διαπραγμάτευση. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα προσέξουμε. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις, θα τα ετοιμάσουμε όλα και θα έχουμε την ευκαιρία για μια συνθετική έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, το υπερθυμόν 12, τη γνωμοδότηση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. Και με μεγάλη μου χαρά δίνω το λόγο στην εισηγητρία Τζουιτ Κέρτιν Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, διότι μπορεί να χρειαστεί να φύγω στις 4 λόγω των ταξιδιωτικών των περιορισμών λόγω του ταξιδιού μου. Αλλά θα σημειώσω όσα θα πείτε. Μπορεί να μην προλάβουμε να τα απαντήσω όλα και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Εμεί συντάξαμε αυτή την γνωμοδότηση προ την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ για την ετήσια έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα του 2015. Και φυσικά όταν μιλάει κανεί για θεμελιώδη δικαιώματα ε, μιλάμε για ένα τεράστιο πεδίο εφαρμογή για την γνωμοδότηση αυτή. Μπορούμε να πούμε ένα σωρό πράγματα για πράγματα που, πήγαν, δεν πήγαν καλά και για κάποια που πήγαν καλά πέρυσι. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε σύντομοι και προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε ε, στην οπτική γωνία της Επιτροπής Αναφορών, δηλαδή τι οι πολίτες βλέπουν ως παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, γιατί αυτό ε, μπορεί να συμβάλλει επικοδομητικά στην έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και έτσι μπορούμε να δώσουμε και φωνή στις ανησυχίες αυτές των πολιτών όπως έχουν ακουστεί εδώ στη δική μας Επιτροπή. Η γνωμοδότηση κατά κύριο λόγο βασίζεται σε αναφορές που έχουμε λάβει μέσα στο 2015. Προσπαθήσαμε να τις συνοψίσουμε και να τις ε, δομήσουμε ε, με τέτοιο τρόπο ώστε να υπογραμμίζονται τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτές τις ε, αναφορές που προκύπτουν από αυτές. Έχουμε λάβει πολλές αναφορές που αναφέρονται στα θεμελιώδη δικαιώματα, πάνω από 100 συγκεκριμένα αναφέρονται στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά αν δει και πολλές από τις υπόλοιπες αναφορές και όταν ε, φτάνουν οι αναφορές στην Επιτροπή συχνά αναφέρονται εμέσως ε, στα θεμελιώδη δικαιώματα λόγω των θεμάτων που αφορούν. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που μπορούμε να καλύψουμε. Κάτι συγκινητικό που είδαμε είναι ότι η ευαισθητοποίηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα έρχεται και από τις τέσσερις γωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βόρο, Νότο, Ανατολή και Δύση. Και ε, οι πολίτες θεωρούν ότι τους αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα υπερασπίζονται πολύ ε, δραστήρια και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ε, η άλλη πλευρά όμως είναι ότι δυστυχώς πολλοί πολίτες αναμένουν από εμάς να μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε απαραίτητα να κάνουμε. Και εκεί υπήρχε ένα κενό μεταξύ των προσδοκιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που υπάρχουν στο χαρτί και είναι πολύ σαφή ε, και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται πραγματικά και χρησιμοποιούνται πρακτικά. Οπότε απομένουν πολλά να γίνουν εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στου πολίτε τι είναι δυνατό σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πότε είναι αναγκαίο να ανελθεί δράση σε εθνικό επίπεδο ή σε άλλα επίπεδα. Γι' αυτό το λόγο υπογραμμίζουμε ήδη από το πρώτο σημείο της γνωμοδότησης αυτή τη συνδέση με το άρθρο 51. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση φέτος με αν θυμάμαι καλά την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ίσως και την ΑΦΚΟ. Σίγουρα ήταν ΛΥΜΠΕ. Και βέβαια αυτό δεν εντάσσεται στο χρονικό πλαίσιο της νομοδότησης, αλλά θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό να κάνουμε αυτή τη σύνδεση με το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Αυτό το άρθρο σύμφωνα με το δικαστήριο επιτρέπει στου πολίτες να απαιτούν συγκεκριμένα δικαιώματα και μπορεί να χρησιμεύσει για ορισμένε υποθέσει και κάποια παραδείγματα θα ήταν η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο το πλαίσιο δραστηριοτήτων της Frontex ε, και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχει, όπως είπα, αυτό το κενό μεταξύ ε, των θεμελιδών δικαιωμάτων και του πώς εφαρμόζονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Ειδικότερα όσον αφορά ζητήματα που αφορούν την ε, ευμερία του παιδιού, το περιβάλλον, την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας και η παροχή ε, υπηρεσιών κοινωνοφιλίας όπως ε, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να ε, περιγράψουμε, να, να προσδιορίσουμε αυτό το κενό ε, ως κάτι πολύ σημαντικό τους γνωμοδότης και κάτι πρέπει να κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω είναι να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο ώστε οι πολίτες να μπορούν να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους και ποιος είναι ο ρόλος των Εθνικών Επιτροπών Αναφορών του Ισδημεσολαβήτριας και των Εθνικών Ομάδων όταν πρόκειται για ζητήματα που είναι εθνικής αρμοδιότητας και όχι ευρωπαϊκής. Πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να δρούν ε, σύμφωνα με το πνεύμα των θεμελιδών δικαιωμάτων ακόμη και αν ε, ενδεχομένως δεν τους δεσμεύει ακριβώς ε, διά, μια συγκεκριμένη διάταξη του χάρτη. Επίσης, ε, επισημαίνουμε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ομάδες αναφορών που αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα όπως τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Είχαμε πολλές αναφορές ε, και για δικαιώματα που σχετίζονται με την ελευθερία κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την άσκηση της ελεύθερης μετακίνησης. Ε, τα πολιτικά δικαιώματα, το δικαίωμα ψήφου, τέτοια ζητήματα σε σχέση με τα δικαιώματα ψήφου. Το είδαμε αυτό με το Brexit. Πολλές τέτοιες αναφορές ήρθαν το 2015 όσον αφορά την ψήφο για το Βρετανικό δημοψήφισμα. Έχουμε ίδια αιτήματα και από άλλε χώρε, όχι μόνο για τη Βρετανία. Η ψηφοφορία στι εθνικέ εκλογέ είναι ένα ζήτημα που έχουμε θέσει στον Επίτροπο ε, Τίμερμαντ ε, πολλέ φορέ. Τα δικαιώματα των ε, ΛΟΑΤ αποτελεί ένα ζήτημα μείζωνο ανησυχία παντού στην Ευρώπη τα δικαιώματα των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα όσον αφορά τη διασυνοριακή κυδαιμονία και τις περιπτώσεις ε, καλής των παιδιών και στις σημερινές συνθήκες με τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προφανώς ε, πολλές αναφορές ε, εκφράζουν ανησυχία για τα δικαιώματα των ετών των άσυλων, των μεταναστών, των προσφύγων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προσπαθούμε λοιπόν να τα παρουσιάσουμε όλα αυτά. Δεν πρόκειται παρά για ένα πλαίσιο ουσιαστικά ως γνωμοδότηση ε, και μέσω αυτής θέλουμε να εκπροσωπούμε τις φωνές ε, των ανθρώπων που έχουν στραφεί εδώ στην Επιτροπή Αναφορών για να τροφοδοτήσουμε το έργο της Επιτροπής ΛΥΜΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τζούντι, κυρία Στανόκα. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την συνάρφο Τζουντ και τον Τάρλινγκ για την πρότασή της που είναι πολύ καλή. Βέβαια, έχω ένα ερώτημα. Και το ερώτημά μου αφορά την ανάγκη Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να προωθούν, ε, να προωθήσουν μάλλον τη γνώση του άρθρου 51 Καλό να το λέει κανείς, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το άρθρο 51 και την εφαρμογή των άλλων άρθρων. Δεν ξέρουμε πως αυτός είναι ένας επιτιδευμένος τρόπος να θέσετε το πρόβλημα το άρθρο 51, αλλά δεν συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει όπως το γράφετε εσείς. Επίσης πολύ καλό είναι το ότι γύρω ορισμένα ζητήματα, για τις αναφορές που λαμβάνουμε, Είχαμε πάει και στο Λονδίνο σε μια διερευνητική επίσκεψη για να δούμε τα προβλήματα που υπήρχαν εκεί με τη μέρη με των παιδιών. Εγώ θα καταθέσω τροπολογίες. Παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά το σημείο 8. γιατί πρέπει να αναφέρουμε και το πρόβλημα της απομάκρυσης των παιδιών από τι οικογένειέ του χωρί την συγκατάθεση των γονέων του. Δεν είναι μόνο δυσυνοριακέ υιοθεσίε. Και από την άλλη πλευρά, ε, με ανησυχεί λίγο κάπω στο σημείο 7, θα καταθέσω τροπολογία από αυτού. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επίκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο το θέμα των ε, συζύγων. Κατά τα λοιπά, είναι ένα πολύ καλά διατυπωμένο κείμενο και νομίζω ότι μπορούμε να το εγκρίνουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Ε, συμφωνώ με πάρα πολλά σημεία της ε, έκθεσης. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και με τροπολογίες να βελτιώσουμε τα θέματα τα οποία έθιξε. Σέβομαι το χρόνο ε, που είναι σύντομος και για την ίδια προκειμένου να παρακολουθεί τη συζήτηση. Επομένως, ε, με αυτή την παρατήρηση ε, ολοκληρώνω την παρέμβασή μου και λέω ότι με τροπολογίες θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τερικαμπράς, παρακαλώ. Όχι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την αγαπητή συνάδελφο για την ε, γνωμοδότηση που είναι δύσκολη διότι πρέπει να καλύψει τόσες πτυχές. Πρέπει όμως να πω κάτι και θα σας εξηγήσω γιατί θα το πω. Νομίζω ότι λείπει η αναφορά στα δικαιώματα των γυναικών. που ε, στην απασχόληση και στην εκπαίδευση δεν έχουν ίση μεταχείριση με τους άντρες. και που υποφέρουν από ε, σεξουαλικές και άλλες επιθέσεις ε, με πολύ σοβαρά αποτελέσματα. υπάρχουν πολλές ε, πράξεις οι οποίες δεν φτάνουν στα αυτιά της Επιτροπής μας, ε, τις οποίες όμως πρέπει να καταδικάσουμε. Με σαφή τρόπο. Η προηγούμενη παρατήρηση για το άρθρο 51 ε, ισχύει και εδώ, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα πριν. Η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν να κάνουν και με πολλές ε, παραβιάσεις που συχνά αναφέρονται στην Επιτροπή μας ε, για θέματα μόλυνσης ε, του περιβάλλοντος κλπ. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν και κάποιες πιο λεπτές, πιο αόρατες πτυχές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διότι συχνά κρύβονται πίσω από πολλές από τις αναφορές που φτάνουν σε εμά. Όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν ε, τον ρατσισμό, το δικαίωμα και η ελευθερία της πληροφόρησης, ε, λογοκρισία και η κατάχρηση εξουσίας. Εάν συμπληρώσουμε στην Επιτροπή μας, αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να καταλάβει ότι ακολουθούμε παρόμοια γραμμή με αυτούς και ότι έχουμε κοινά προβλήματα και συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα ο Πάλ, τέλος. Ε, ευχαριστώ πολύ Σεσίλια. Βέβαια, η κυρία Μετσόλα είναι αρμόδια για το θέμα αυτό από πλευρά ΣΕΛΚ. Δεν μπορούσε όμως να παραστεί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων σήμερα. Και εδώ έχω μπροστά μου γραπτός την δική της ε, άποψη. Θα σας πω λοιπόν τι γράφει εδώ. Χαιρετίζουμε ως ομάδα το σχέδιο γνωμοδότησης. Έχουμε ανισχύσει για κάποια θέματα του κειμένου, ιδίω εκεί που αναφέρεται η Frontex. κυρία Μετσόλα λοιπόν θεωρεί ότι το κείμενο σχετικά με τη Frontex θα πρέπει να είναι στο δυνατόν πιο κοντά σε αυτά που περιλαμβάνονται στην έκθεση ΛΥΜΠΕ ε, για τη Frontex, μια έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας, την οποία στήριξαν περισσότερες πολιτικές ομάδες και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Έχει καταθέσει τροπολογίες, κυρία Μετσόλα, ώστε να σχετιστεί ε, και να αναφέρεται, μάλλον να συνάδει με το χάρτη η έκθεση. Πάντως ό,τι αφορά το θεμελιώδης δικαίωμα στην περιβαλλοντική προστασία και άλλα ε, μας βρίσκουν σύμφωνο. Σε ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Εύη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο για το έργο της. Ε, με βρίσκει σύμφωνη. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που θα ήθελα να προσθέσουμε οποίο μου φαίνεται ότι σχετίζεται με αυτό που περιγραφεί η συγκέντρια στην παραγραφό 1. Ναι, αλήθεια, έχουμε τι προσδοκίε των πολιτών για την προστασία των συμπολιτών του δικαιωμάτων, οι οποίε ε, τη χάνουν απογοήτευση διαρκώς. Ένας από του λόγου αυτής τη απογοήτευση, κατά την απόψή μου, είναι η κοινική και διαρκής εφαρμογή σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό των μέτρων λιτότητας τα οποία ακόμα υιοθετούνται ως ε, ε, οικονομική προσέγγιση αναφοράς ε, και που δεν δίνει αποτελεσματικές απαντήσεις αλλά οδηγεί σε μια δραματική κατάσταση 8 χρόνια μετά από την αρχή της κρίσης όπου συνεχίζουμε να παρατηρούμε επιδίνωση των επιπέδων φτώχειας υψηλών ποσοστών ανεργίας ανήκουστων και αβεβαιότητα κυρίως μεταξύ των νέων. Αυτές ε, είναι οι αιτίες που κατά την απόψή μου ε, πρέπει να προσθεθούν και θα, εγώ θα υποβάλω τις σχετικές τροπολογίες ώστε να κάνουμε τι, να προσπαθήσουμε πολιτικά να το φωνάξουμε δυνατά και καθαρά ότι χρειάζεται να αλλάξουμε ρότα, να δείξουμε υπευθυνότητα. Προς τον πλησίον μας φυσικά ε, αυτό έπρεπε να ισχύει ήδη, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, οπότε κατά την απόψή μου πρέπει να προταθούν αυτές οι τροπολογίες ώστε να εμπλουτίσουμε ε, ε, λίγα λόγια βέβαια που επιτρεπόταν να αναφερθούν σε αυτή την έκθεση όπως η προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων όπου φυσικά όλοι μας ε, δείχνουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτήν την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank you, Eleonora. Now we... Σε Έχουμε και εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θέλετε το λόγο, όχι. Α, εντάξει. Τότε, εσείς κυρία Κίρτον Τράλινγκ, θέλω να προσθέσετε κάτι ή... Θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφους για τα σχόλια και περιμένω με ανυπομονησία και τι τροπολογίε. Όπως είπα και στην αρχή, εμείς συστηθήκαμε σε αυτό που λέει η αναφορά και τι θα θέλαμε να είχαμε πάρει δεν πήραμε. Υπάρχουν βέβαια θεμητέ ανησυχίε. Ακούσαμε τον κύριο Τερικάμπρα, δικαιώματα των γυναικών. Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν πήραμε πολλέ αναφορέ. Άρα εμείς έχουμε περιοριστεί σε αυτά που ανέφεραν οι αναφορές. Αν υπάρχουν και άλλα θέματα, ναι, και φυσικά μας ενδιαφέρουν και αυτά, αλλά με τα χαράς να λάβω και υπόψη την ε, προοπτική της ΛΥΜΠΕ. Περιμένω τις τροπολογίες σας τώρα και ελπίζω με βάση και τις συμβιβαστικέ ε, να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση. Με βάση και την προηγούμενη εμπειρία μου είμαι βέβαιη ότι θα λάβω πολλές τροπολογίες. Λίγη υπομονή, λίγη ανοχή λοιπόν ζητώ από όλες τις πολιτικές ομάδες για να καταλήξουμε σε μια καλή συμβιβαστική νομοδότηση που θα μπορέσει να ψηφιστεί μετά. Βεβαίω, είμαι πεπισμένη ότι θα το πράξετε αυτό, λέει η πρόεδρο, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, 15 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Άρα δεν έχετε αρχέ να συντάσσετε τι τροπολογίε, ξεκινήστε τάχιστα. Και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μα θα λάβει χώρα στι 11 Οκτωβρίου. Τα καταφέρατε και μείναν και δύο λεπτά για να προλάβετε. Πάρτε ανάσα και συνεχίστε τον αγώνα. Και τώρα προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, πρόκειται για το σημείο 13. Ε, αναφορά υπαριθμών 1196-0650 και την αναφορά υπαριθμών 0207 για τη γλυφοσάτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τρεις αναφέροντες ε, τρεις αναφορές που μπορούμε να εξετάσουμε ταυτόχρονα, διότι έτσι μπορούμε να έχουμε οριζόντια προσέγγιση. Οι αναφέροντες δεν είναι εδώ, είναι όμως ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Φόλκερ Βάφλετ και του δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή εδώ συζητάει τρεις αναφορές και οι τρει ζητούν απαγόρευση τη γλυφωσάτη, του φυτοφαρμάκου γλυφωσάτη. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της ανθρώπινης ε, της ε, υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος και παραπέμπουν σε μελέτες που δείχνουν κατά τη γνώμη τους ε, τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης της γλυφοσάτης ε, στα φυτοφάρμακα. Η Επιτροπή ήδη έχει απαντήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε αυτές τις αναφορές και θα ήθελα να συνοψίσω τα βασικά σημεία. Η γλυφοσάτη πρόσφατα εξετάστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πιθανή ανανέωση της έγκρισής της για την ε, αξιολόγηση αυτήν ε, ήταν διαθέσιμος ε, ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός μελετών, πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που βλέπουμε συνήθως για τέτοιες ουσίες. Μερικές ήταν κάποιες που παρουσίαζαν κατευθείαν γραμμές, άλλες ήταν επιστημονικές μελέτες με αναθεώρηση ομοτήμων. Κάποιες ήταν ε, γερμανικές, ε, τις οποίες ε, μετά αξιολόγησαν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, καθώς και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η ΕΦΣΑ. Έτσι είχαμε μια πολύ σφαιρική και αξιόπιστη αξιολόγηση, η οποία συνοψίζεται στα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ και το, τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ για τη γλυφοσάτη ε, δείχνουν ότι υπάρχουν ασφαλείς χρήσεις για τη γλυφοσάτη σε φυτοφάρμακα. Ασφαλής χρήση σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προϊόν ε, χωρίς αρνητικές συνέπειες ε, για τους ανθρώπους και τα ζώα και χωρίς απαράδεκτα αποτελέσματα για το περιβάλλον. Υπό το φως λοιπόν αυτής ε, της ευνοϊκής αξιολόγησης ε, της ΕΦΣΑ, η Κομισιόν δεν έχει λόγους να απαγορεύσει τη γλυφοσάτη. Αυτή τη θέση φαίνεται να συμμερίζεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να θυμάστε ότι φέτος τον Απρίλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα όπου καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανανεώσει την έγκριση της γλυφοσάτης για ε, περιορισμένο χρονικό διάστημα, 7 χρόνια. παρόλα αυτά όμως δόθηκε ε, έγκριση, μάλλον ε, υποβλήθηκε αίτημα για ανανέωση της άδεια για την γλυφοσάτη. Δύο από τις αναφορές που εξετάζουμε είναι από προηγούμενες χρονιές και τον τελευταίο μήνα πριν τις θερινές διακοπές είχαμε νέες εξελίξεις στο θέμα αυτό και γι' αυτό θα ήθελα να σας περιγράψω την κατάσταση σχετικά με το τι συνέβη σε αυτούς τους μήνες. Μπορεί να γνωρίζετε ότι τα κράτη-μέλη δεν κατέληξαν σε απόφαση σχετικά με την παράταση της έγκρισης της γλυφοσάτης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον έπρεπε να λάβει απόφαση, αποφάσισε να παρατείνει την άδεια της γλυφοσάτης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι δηλαδή η ΕΧΑ, ο Οργανισμός ε, Χημικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκδώσει γνωμοδότηση για την ε, ταξινόμηση της λιφωσάτη και το αργότερο μέχρι το τέλος του 2017. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει στα κράτη-μέλη ένα δεύτερο κείμενο να περιοριστούν οι προϋποθέσεις χρήσης της λιφοσάτης ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτές οι περιορισμένες προϋποθέσεις εγκρίθηκαν από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Αυγούστου. Αυτοί οι επιπλέον περιορισμοί περιλαμβάνουν απαγόρευση μιας ε, σύνθεσης ε, που βασίζεται στην γλυφοσάτη, συμπεριλαμβάνουν την ε, υποχρέωση να εξετάζεται πιο προσεκτικά η χρήση πριν τη συγκομιδή και επίσης η περιορισμένη χρήση σε ε, ε, δημόσιους χώρους όπως είναι τα πάρκα ή οι παιδικές χαρές. Αυτά είναι σύντομα τα πιο πρόσφατα γεγονότα στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια ουσία την οποία συζητούν όλοι αυτές τις μέρες. Τώρα λοιπόν που θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές. Νομίζω ότι θα συζητήσουμε αρκετά το θέμα αυτό. Παρακαλώ λοιπόν συγκεντρωθείτε και να, είμαστε, να παραμείνουμε εντός θέματος. Ελεονόρα, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Θεωρώ ότι για το ζήτημα της γλυφωσάτης ε, είναι αναγκαίο να μην αποδυναμωθεί η προσοχή. Γι' αυτό το λόγο οι αναφορές πρέπει να μείνουν ανοιχτές. Το λέω αυτό πρώτο-πρώτο εισαγωγικά, διότι τα όσα μόλις μας ανέφερε η Κομισιόν πολύ σωστά μας ε, υποδεικνύουν ποια ε, είναι τα μελλοντικά δρόμενα, τα μελλοντικά σενάρια. περιμένουμε του χρόνου τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Χημικών Ουσιών που θα δώσει την απάντησή της για την επιστημονική αξιολόγηση αυτού του φυτοφαρμάκου. Και η ολόκληρη ιστορία που έχει προηγηθεί είναι γεμάτη εμπόδια. Κατά την απόψη μου η είναι ένα ισχυρότατο φυτοφάρμακο το οποίο θα πρέπει να απαγορευτεί το συντομότερο δυνατόν. Τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί ε, προσωρινή ανανέωση είναι σαφές ότι κατά κάποιο τρόπο να έχουν καθορίσει την κατάσταση. Πολλά όμω θα πρέπει να αξιολογηθούν. Εγώ θεωρώ ότι το να διατηρήσουμε ανοιχτέ αυτέ τι αναφορέ θα αποτελέσει ακόμα ένα κίνητρο ώστε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Το πραγματικό πρόβλημα, το πραγματικό ζήτημα επί της ουσίας είναι μια μετάβαση σε ένα διαφορετικό γεωργικό μοντέλο που δεν θα χαρακτηρίζεται από τη μεγιστοποίηση του κέρδους ε, και από τη βιομηχανική γεωργία η οποία χρησιμοποιεί τέτοιου είδους ουσίες οι οποίες να θυμίσω συμβαδίζουν με τα μεταλλαγμένα υπενθυμίζω και με έναν άλλο τύπο γεωργίας που δεν χρειάζεται η Ευρώπη κατά την άποψή μου οπότε είναι ευπρόσδεκτες τέτοιου είδους αναφορές που ευαισθητοποιούν το κοινοβούλιο όσον αφορά ε, το τι γίνεται στο έδαφος ε, ε, διότι πολλοί γεωργοί επιμένουν και απαιτούν μετάβαση προς μια γεωργία πιο βιώσιμη και εφόρο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τερικαμπράς. Ευχαριστώ πολύ. Η ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλισης των Τροφίμων, είναι μια πραγματική αρχή, όπως λέει το όνομά της και αναφέρεται, αναφέρθηκε από το Κομισιόν ε, όλη την ώρα ε, αυτό, αυτή η αρχή. Αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις και άλλες νομοδοτήσεις. ακόμα και η ΕΦΣΑ, ξέρετε, δεν έχει καταλήξει σε κάτι σε όλα τα σημεία. Για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Πρώτον, για το θέμα της, ε, των βλαβών προς την υγεία, ε, ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας ε, του Καρκίνου ε, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη είναι πιθανός ε, καρκινογόνος στους ανθρώπους. Διάφορες μελέτες δείχνουν επίσης ότι τα φυτοφάρμακα που περιλαμβάνουν ενδοκρινικούς διαταράκτες δημιουργούν χάος στις ορμόνες και μπορούν να επηρεάσουν τη γονιμότητα. Δεύτερον, εάν διοπιστωθεί μακροχρόνιος κίνδυνος για τα ζώα, όπως και για τα ζώα ακροκτήματων, όπως, της όπω όπως ε, τα πρόβατα, και οι Αγελάδες ε, και η σχετική Γερμανή αρχή έχει βρει επιπτώσεις για τη βιοπικιλότητα ε, λόγω των λοιπασμάτων γενικότερα και πιο συγκεκριμένα της γλυφοσάτης. Τρίτον, τα μεταλλαγμένα και η γλυφωσάτη είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Τέταρτον, η αντίσταση στην γλυφοσάτη, η οποία είναι δεδομένη ήδη στην ΙΠΑ και στον Καναδά, ε, είναι διαδεδομένη λόγω των, ε, της χρήσης των μεταλλαγμένων ε, και τα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με την ΕΦΣΑ ε, λένε ότι υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο όπου 8 από τις 24 ετούντες ε, συμπεριλαμβανομένες της Μονσάντο παρουσίασαν τα στοιχεία για την γλυφοσάτη που δεν υποστηρίζονται από την ψυχολογική αξιολόγηση έκτον έλλειψη διαφάνειας. Τα συμπεράσματα της έκθεσης της ΕΦΣΑ όσον αφορά ε, το καρκινογόνο χαρακτήρα της γλυφοσάτης βασίζονται στα στοιχεία κάποιων δημοσίευτων μελετών της, του ίδιου τομέα. Και εβδόμων υπάρχουν εναλλακτικέ. Οι βιολογικοί καλλιεργητές έχουν αποδείξει το έχουν αποδείξει ξανά και ξανά ότι η γλυφοσάτη δεν είναι αναγκαία για ε, τη υψηλή παραγωγικότητα της γεωργίας. Η γεωργία του μέλλοντος ε, συνεργάζεται με τη φύση και όχι κατά της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει το λόγο. Α, όχι. Ξέχασα. Κύριε Σακοράφ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μόνο για μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι και δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω. Αυτό που θέλω να έχουμε στο νου μας, επειδή ακριβώς παίρνουμε αποφάσεις εμείς εδώ, είναι ότι Πρόκειται για ένα ισχυρό δηλητήριο. Αυτό είναι παραδεκτό από όλου, όπω είπατε και εσεί, ε, συζητιέται πάρα πολύ αυτόν τον καιρό. Είναι κάτι που μπορεί να το χρησιμοποιούμε και εμεί, μπορεί να το χρησιμοποιούν τα παιδιά μα, ε, να το προσλαμβάνουμε. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μα, ότι δεν μιλάμε μόνο για κάποιου που δεν μα αφορά το θέμα, μιλάμε και για μα. Άρα πρέπει, κατά τη δική μου άποψη, να την κρατήσετε ανοιχτή αυτή την υπόθεση και όπω είπαν και οι συνάδελφοι, να την παρακολουθούμε επισταμένα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ευχαριστώ ευχαριστώ. Okay, so let me then now try to... Ας προσπαθήσω να συνοψίσω. Όπως είπε και η κυρία Κοράφα, θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς ε, το, ζήτημα αυτό και φυσικά και θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Και επειδή μόλις τον Ιούλιο στήριξα τα κράτη-μέλη μια πρόταση για να τεθούν ε, όρια στην χρήση του ζανιοκτώνου γλυφοσάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπατε όμως και όλοι σας. Έχουμε ε, ουσιαστικά ατάκτως ερημένα στοιχεία από εδώ και από εκεί. Υπάρχει το 18μηνο. Όταν περάσει μπορεί να υπάρξει μια νέα συζήτηση και μια νέα αξιολόγηση. Το θέμα όμως ακόμη είναι ανοιχτό. Δεν ελήφθη τελική απόφαση. Άρα είμαστε κάπως, ε, θα έλεγα, σε μεταβατική περίοδο. Οπότε αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και παραμένουμε σε επαφή με την Κομισιόν. Και σε 1,5 χρόνο τα ξαναλέμε. Ωραία. Λοιπόν, επόμενη αναφορά 1338 το 2012 Μαρκ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά των Νεολικών Πάρκων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις Πηγέ Πηγές Ενέργειας. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο, τον κύριο Πάρκ Φόρμπς. Ευχαριστώ πολύ η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά των Ολικών Πάρκων έχει οργανώσεις από 31 χώρες, 250 είναι σαφείς οι, ε, ε, οι απόψεις μας. Στόχος ήταν ε, η πολιτική της να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αλλά και να γίνει σεβαστό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε συμφωνίες. Αν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ σύμβασης ε, και των οδηγιών, όπως είμαστε στο άλλο παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να εφαρμόζεται οι συνθήκες και όχι το δευτερογενές δίκαιο. Έχετε παρουσίαση, έχετε μια αναλυτική έκθεση. Σας ενημερώσαμε και τον Ιούνιο ότι οκτώ κράτη-μέλη και η Ένωση είναι στον κατάλογο των μη συμμορφώνων ε, συμβαλωμένων μερών. 5-9G είναι απόφαση για τη μη συμμόρφωση. Δεν έχει το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο η Ένωση. Ούτε σαφεί οδηγίε δίνει ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν σωστά τι απαιτήσει τη σύμβαση για τη δημόσια συμμετοχή οι χώρε μέλη. Σε ό,τι αφορά τα σχέδια δράση για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. 20% ανανεώσιμε πηγέ μέχρι το 2020. Αυτό λέει η συνθήκη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση, δεν έχει ε, παρακολουθεί επαρκώς η χάρη είναι ένα παράδειγμα. Η οδηγία λοιπόν έχει νομικά κενά και σφάλματα. Δεν είναι διαφανής, δεν είναι δίκαιης, δεν δίνει πληροφορίες ε, στην κοινή γνώμη στους πολίτες. Δεν μπορεί ε, το κοινό να συμμετέχει, δεν υπάρχει δημόσια συμμετοχή δεν εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται υπόψη ε, η έκβαση της δημόσιας συμμετοχής. Ε, τον Οκτώβριο θα έχουμε τη δεύτερη έκθεση πρόοδου της γιούρνησης. Στην πρώτη λέει ότι η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τότε δραστηριότητες ε, δεν ήταν επαρκείς για να αντιμετωπίσουν τις συστάσεις, δεν προβλέπουν κανένα σχέδιο δράσης, κατάλογο προτινών δραστηριοτήτων, ούτε και εξηγούν το πώς προτείνεται το μέρος να εφαρμόσει τις συστάσεις. Άρα θεωρεί η Επιτροπή ότι το λόγο δεν πληρεί τις απαιτήσει της απόφασης 79G. Ε, ε, Ούτε έχει κάνει κάποιο προ αυτή την κατεύθυνση. Να σα πω ότι η σύμβαση του Άρχου απαιτεί την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών, αλλά πάει πιο πέρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ζητάει πιο αναλυτικέ εκτιμήσει, στατικέ εκτιμήσει περιβαλλοντικού αντικτύπου. Στο Journal of Energy and Natural Resources ε, Law δημοσιοποιήθηκε ένα άρθρο, βλέπετε τον τίτλο του, στη διαφάνεια και μιλά για τις, ε, ε, πέτοι περίπτωση της Ιρλανδίας και τα ολικά αυτά πάρκα. Υπάρχει ε, νομολογία. Η απόφαση Σόρτς από τη Γεννήση δείχνει ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στην πολιτική της Ιρλανδίας ό,τι αφορά την ολική ενέργεια. η αγορά είναι άκρος ασταθής και υπάρχει κίνδυνος ε, από τέτοιου είδους επενδύσεις, ότι γνωρίζουμε για το κόστος, τα ωφέλη, τον αντίκτυπο, μέτρα μετριασμού κτλ. κτλ. Αν δούμε το 5-3 του υποδείγματο τη ΡΕΑΠ, που το έχουν αφήσει και ενώ 19 από τα 27 κράτη-μέλη δεν έχουν δώσει ε, άλλα δε ε, επαρκείς πληροφορίες Βλέπουμε και τι λέει και ο Επίτροπο Ενέργεια. Δεν θέλουμε λοιπόν να, έχουμε έναν υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τα κράτη-μέλη. Τι θα γίνει με τι ανανεώσιμε πηγέ, Πώ θα μειώσουμε τι εκπομπέ θερμοκηπιακών αερίων κτλ. κτλ. Τώρα, ε, βλέπουμε ότι πρόκειται για πραγματική φάρσα ε, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό. Έχουμε εξοικονομήσει σε ό,τι αφορά εκπομπέ ε, διοξιδίου του άνθρακα υπάρχουν παράγοντες που δεν μπορούν να προκαθοριστούν σε ό,τι αφορά το πώς θα επηρεάσει ε, ή θα μειώσει τα θερμοκηπιακά αέρια αυτή η πρόταση. Δεν αιτιολογείται από μόνο του αυτό το σχέδιο ότι θα οδηγήσει στη μείωση των θερμοκηπιακών αερίων. Θα δικαιολογηθεί μόνο αν φανεί ότι συμμορφούνται προ τι γενικέ δημόσιε πολιτικέ για τη μείωση των, των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων. Άρα τελικά σπαταλούμε ένα τρία, ένα τρεις ευρώ για τις ανεμογεννήτριες, για τα φωτοβολταϊκά. Τι λέει ο Ζαν Φρανσουά Μπρέικλαντ από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Περιβάλλον και επικεφάλης ομάδας Α2. Λέει ότι αν αντί μίας ε, 110 μέτρων ε, είχαμε ένα ε, μεταλλικό άγαλμα του Μίκη Μάους 110 μέτρων ε, θα κοιτάζαμε την, ε, το ισοζύγιο άνθρακα. Γιατί το κοιτάμε στην προκειμένη περίπτωση. Άρα τι βλέπουμε να υπάρχουν δυσλειτουργικές πολιτικές. Είναι η Ιρλανδία παγκοσμίω γνωστή για την κληρονομιά της. Πώς λοιπόν τολμούν, αφού το περιβάλλον της Ιρλανδίας ανήκει στις πολίτες της χώρας, πώς μπορούν κάποιοι να προωθούν ένα τέτοια δυσλειτουργικό σχέδιο που θα καταστρέψει το μοναδικό αυτό τοπίο με τεράστιες γιγαντιές τουρμπίνε και κάτι που είναι παράνομο και καταχρότητα των δικαιωμάτων. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον Αγγέλη Χερέρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον αναφέροντα για την σαφή παρουσίαση του. Ισχυρίζεται ότι η πολιτική για τις ανεμογεννήτριες ε, αντίκειται στην ε, στην ε, σύμβαση του Όρκους. Το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει την συμμόρφωση των κρατών μελών με την ε, σύμβαση του Όρκους. Όσον αφορά τα ευρήματα και τις συστάσεις της Επιτροπής Συμμόρφωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει επιστολές προς όλα τα κράτη-μέλη και τα ενημερώνει για τα ευρήματα και τους θυμίζει ότι πρέπει να σέβονται τις ρήτρες της σύμβασης ε, του όρχους. Και ε, εφόσον είναι απαραίτητο θα πρέπει να υποβάλουν αναθεωρημένο ε, σχέδιο δράσης. Η ε, Κροατία, για παράδειγμα, νέος κράτος μέλος έπρεπε ε, να υποβάλει σχέδια κατά την προσχώρησή της. Και επίσης τα κράτη-μέλη πρέπει στην έκθεση πρόοδου που υποβάλλουν κάθε δύο χρόνια να συμπεριλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των μέτρων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σύμβασης. Ε, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αξιολογούν αυτή τη στιγμή τις απαντήσεις των κρατών μελών και θα ζητήσουν περισσότερα στοιχεία από κράτη-μέλη εφόσον διαπιστώσουν ότι δεν είναι ικανοποιητικές, ε, απόλυτα ικανοποιητικές οι απαντήσεις τους. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η πρώτη αναθεώρηση της Επιτροπής συμμόρφωση στην οποία αναφέρθηκε και ο αναφέρον βασίζεται σε μια ήδη πεπαλαιωμένη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, του 2014. Δεύτερη έκθεση υπέβαλε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015, την οποία θα εξετάσει η Επιτροπή Συμμόρφωσης ε, φέτος τον Οκτώβριο και μέχρι φέτος τον Οκτώβριο και η τρίτη ε, έκθεση πρόοδου θα αποσταλεί εντός του έτους. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τις ε, απαιτήσεις της Σύμβασης του Όρχους ε, κατά την εκπόνηση της ε, επικείμενης νομοθετικής πρότασης. Ο αναφέρον επίσης ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα ωφέλη των επενδύσεων Στι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Ωστόσο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ενέργειας σε, σε τακτική βάση υποβάλλει εκθέσει σχετικά με τι εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Στην έκθεση του 2016 επισημαίνει ότι... Ε, αποφύγαμε 380 εκατομμύρια τόνους ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, για να καταλάβετε τι αντιπροσωπεύει το νούμερο αυτό ε, καλύπτει τις επομπές αερίων του θερμοκηπίου της Πολωνίας σε ένα χρόνο. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών ε, με διαφορετική μεθοδολογία έχει καταλήξει σε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. έχουμε εξοικονομήσει, υπολογίζεται το 1 τρίτο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, και συνολικά το ίμιση των εκπομπών ε, στον τομέα του ηλεκτρισμού. Η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει κατά 110 ε, εκατομμύρια ε, ε, ισοδύναμους τόνους πετρελαίου το 2015, δηλαδή το συνολικά το 10% της συνολικής κατανάλωσης σε ορυκτά καύσιμα. Αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έτσι έχουμε εξοικονομήσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014 λόγω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με έκθεση του 2014 έχει αυξηθεί η απασχόληση με ε, μισό εκατομμύριο πρόσθετες θέσεις εργασίας από το 2008 μέχρι το 2014 λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 1,11 εκατομμύρια εργαζόμενους απασχολεί ο τομέα ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και η μεγαλύτερη αύξηση είναι στι ανεμογεννήτριε. Η σχετική βιομηχανία. Ε, σημαίνει ότι ε, μεταξύ των έξι εταιριών με τις μεγαλύτερες πωλήσει σε ανεμογεννήτριες, οι τέσσερις ήταν ευρωπαϊκές το 2012. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φεραίρε. Εξαιρετικά νέα αυτά υπάρχουν ε, νέε ευκαιρίε απασχόλησης για τόσους Ευρωπαίου πολίτες. Αυτά είναι πολύ καλά νέα. Γιάρα και έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Πιστεύω ότι πρέπει να την κλείσουμε αυτή την αναφορά. Να την κλείσουμε πιστεύω διότι αντιπροσωπεύει την ιδέα το ότι είναι κατά των ε, αιωλικών πάρκων. Τη σέβομαι αυτή την άποψη, δεν την ε, ασπάζομαι όμως. Πιστεύω όμως ότι ε, ε, ε, εντάξει καταλαβαίνω ότι είναι από τη Γαλλία ο αναφέρον και αν πιστεύει ότι δεν πρέπει να στηθούν τέτοια αιωλικά παρκά στη Γαλλία ας το αναφέρει στις τοπικές εθνικές αρχές. Αλλά θα προτιμούσα να μην πήγε στη δική μου αυλή. Είμαι πεπισμένος ε, ότι η κυβέρνησή μου και οι αρχές της Πολωνίας κάνουν ό,τι μπορούν ώστε αυτά τα αιωλικά πάρκα να μην τοποθετηθούν σε ε, μέρη όπου δεν θα έπρεπε να τοποθετηθούν. Καταλαβαίνω τον αναφέροντα, ο οποίος είναι κατά των αιωλικών αυτών πάρκων, αλλά προ τα εκεί κινούμαστε για το μέλλον, για την παραγωγή ενέργεια και αν κάνουμε σωστά τα πράγματα, έχοντα υπόψη μας και λαμβάνοντα υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να στηθούν τέτοια ολικά πάρκα στα κράτη-μέλη, τα οποία επιθυμούν να τα έχουν στο εδάφη του. Για άλλη μια φορά λοιπόν προτείνω να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Κυρία Σακουράφα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να καταργηθούν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην αιωλική ενέργεια όπως ζητάει ο αναφέρον. Πιστεύω όμως ότι είναι χρέος μας να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε αυτά τα προγράμματα. Θέλω λοιπόν να επισημάνω με αυτή την ευκαιρία τα εξή ότι ο αναφέρον καταγγέλει την παραβίαση της συνθήκης άρχους, ε, πράγμα που δεν αντιμετωπίζουμε όπως οι περισσότεροι ξέρουμε εδώ μέσα για πρώτη φορά. Στην απάντησή της η Επιτροπή μας διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της συνθήκης. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι σε προσωπικές επαφές με αναφέροντες πολλές φορές μου έχει καταγγελθεί ότι υπάρχει αυτή η παραβίαση και πολλές φορές η διαδικασία έπεται της απόφασης ή αν γίνεται γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή κατά την άποψή μου να εξετάζει διεξοδικότερα σε κάθε αναφορά που μας γίνεται αν οι διαδικασίες γίνονται, αν είναι ουσιαστικές και αν πληρούν τελικά το σκοπό για τον οποίο γίνονται. Έτσι που οι πολίτες να μην έχουν όλη την πληροφόρηση, όπως και πρέπει εξαιτία της συνθήκης, αλλά και ουσιαστικά να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Στη συγκεκριμένη αναφορά, ο διομασολαβητής ζήτησε να ληφθούν υπόψη ορισμένα έγγραφα. Στην απάντησή της η Επιτροπή μας ενημερώνει ότι δεν προέβησε ενέργεια σχετικά με αυτά τα θέματα. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή, κατά τη δική μου άποψη, να αιτιολογεί αναλυτικά και επαρκώ του λόγου που δεν προέβη σε παραπέρα ενέργειες, ώστε και εμείς αμέλη της Επιτροπής, αλλά και πρωτίστως αναφέρον, να είμαστε βέβαιοι και οι δύο πλευρέ δηλαδή, ότι το θέμα διαρευνήθηκε διεξοδικά. Γι' αυτό θα έλεγα, κυρία Πρόεδρε, επειδή ακριβώ αναφέρθηκε προηγουμένω από την υπεύθυνη ότι η Κομισιόν βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγηση των απαντήσεων των κρατών μελών, να παραμείνει ανοιχτή η υπόθεση, ώστε να μπορούμε να έχουμε την ενημέρωση για το θέμα αυτό και στο μέλλον. Αυτά και σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στερικάβρας. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Μιλώ ως μέλος των Πρασίνων και κατά την άποψή μας τα υπαρκτά στοιχεία και οι προοπτικές ε, μιλούν κατά της έκθεσης του αναφέροντος οπότε πλέον ε, προτείνω να την κλείσουμε την αναφορά αυτή okay. Nobody... Ωραία Κανείς άλλος δεν έχει ζητήσει το λόγο Προτείνω λοιπόν να κάνουμε ακριβώς αυτό, να κλείσουμε την αναφορά. Ε, είχαμε παρόμοιες αναφορές ε, που μας απασχόλησαν και σήμερα το πρωί και πιστεύω ότι η πολιτική βούληση της παρουσίας επιτροπής είναι να επικυρώσει τη σπουδαιότητα μιας μετάβασης από την ορεκτή ενέργεια στην ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και από εκεί πέρα είναι εθνική αρμοδιότητα το να αποφασιστεί αν θα τοποθετηθούν νεολικά πάρκα ανεμογεννήτριες ε, ποιο θα είναι το ενεργειακό μείγμα της εκάστοτε χώρας. Ε, δεν πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να παρεύουμε εμείς υπερβολικά σε κάτι τέτοιο. Προτείνω λοιπόν να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Would, the petitioner like to comment Θα ήθελε να αναφέρον να σχολιάσει. Your beliefs are your beliefs. Αυτό που πιστεύετε είναι δικό σας πιστεύω. Αν εσείς πηγαίνετε και επιβάλλετε τα πιστεύω σας σε άλλους ανθρώπους με μια επίσημη συνένωση χωρίς ανάλυση θα υπάρξει, θα σας έρθει μπούμεραγκ. Ξέρετε, μπορούμε και να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε, αλλά κλείνουμε την αναφορά αυτήν. Και περνάμε στο επόμενο σημείο το 15, το οποίο ήδη συζητήθηκε το πρωί, το 16 ε, επίση και περνάμε στο σημείο 17 αναφορά 1064 του 2011 αφορά την ύπαρξη στρατηγικής ε, εκτίμηση αντικτύπου για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην Εξτραμαδούρα. Ο Ζήλ Σουσό ε, εκπροσωπεί τον ε, αναφέροντα. Do I have the, uh, Do I speak now? Ναι, να μιλήσω τώρα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ ω μέλο την Ενεργία Πατριμόνια Εθνάλ Κουλτουράλ στα Μαδούρα φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Εστρεμαδούρα μεταφράζεται αυτό. Αυτό προσπαθούμε να προστατεύσουμε, αυτή την κληρονομιά προσπαθούμε να προστατεύσουμε και σε αυτήν την ε, αναφορά καταγγέλουμε την ε, παραβίαση του 242 το 2001 για τις μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου σχέδιων και προγραμμάτων. Στην Ισπανία έχουμε 18.000 ανεμογεννήτριες αλλά ποτέ δεν έγινε μία στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, SEA. Αυτό συνιστά κατάφορη παραβίαση και της σύμβασης ε, του Άρχους και της, οδη, της Οδηγίας 42-2001. Μεταφράζω από τα Ισπανικά τώρα. Έχουμε την Ορνηφολογική Εταιρεία της Ισπανίας, η οποία αφού εξέτασε 136 εκθέσεις προόδου και αντικτύπου των ανεμογεννητριών των ολικών πάρκων ε, στη, στα πτηνά στην Ισπανία. 6 με 18 εκατομμύρια πτηνά ε, και με νυχτερίδες ε, μεταξύ αυτών θανατώνονται από τις ανεμογεννήτρες κάθε χρόνο. Σημαντικότερη μελέτη που έχει γίνει ποτέ από ορνηθολογική εταιρεία. Η Στραμαδούρα που είναι μια αυτόν περιφέρεια με δική της κυβέρνηση στην Ισπανία δεν έχει μέχρι στιγμής ε, ανεμογέννητρε γιατί έχει λίγο αέρα γενικά με τη συμβατική ενέργεια παράγει τετραπλάσια ενέργεια από αυτή που καταναλώνει. Άρα δεν χρειάζεται περισσότερη ενέργεια. Όμως η κυβέρνηση τη Στρεμαδούρα θέλει ανεμογεννήτριες πώς να το πω γιατί τις θέλει τώρα είναι αμφίβολο ο λόγο για του οποίου τις θέλει αυτές τι ανεμογεννήτριες η κυβέρνηση στην Εστρεμαδρόπο. όπω είπα δεν έχει και πολύ αέρα, Όμω έχει καλές σχέσει με πολλά λόμπι και κερδοσκόπους στην ενέργεια. Αυτές οι περιστρεφόμενες πόρτες μπαίνουν από τη μια στην διοίκηση ε, και οι διοίκηση βγαίνουν από, ε, άνθρωποι της διοίκησης βγαίνουν από εκεί και βρίσκουν δουλειά σε επιχειρήσεις που κερδοσκοπούν με τον αέρα, με την αιωλική ενέργεια ακόμη και σε περιοχές όπως την Εστρεμαδόρα που δεν φυσάει. Η κυβέρνηση της Εστρεμαδούρα δεν έχει σχέδιο επί της ουσίας για όλες αυτές τις ανομογέννητες που θέλει να εγκαταστήσει. Και βέβαια δεν έχει ούτε εκπονήσει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Και αυτό είναι σκόπιμο, γιατί δεν θέλει να κάνει αυτή τη μελέτη, γι' αυτό και δεν έχει κάποιο σχέδιο. Όπως θα έπρεπε να ε, κάνει, γιατί αυτό απαιτείται από την οδηγία και από τη σεβαστό άρχος, το να γίνει αυτή η μελέτη αντικτύπου. Προσπαθεί λοιπόν να αποφύγει τη διεξαγωγή αυτή τη μελέτη. Και έτσι ούτε καν σχέδιο δεν έχει φτιάξει. Άρα οι εργολάβοι μελετούν το χάρτη της Εστρεμαδούρα και επιλέγουν αλακάρτ. Εδώ θα φτιάξουν ελικό πάρκο, εκεί θα φτιάξω άλλο ένα και επηρεάζουν ε, κάποιους μέσα στην κυβέρνηση και έτσι γκρίνονται αυτά τα ε, αιωλικά πάρκα, χωρίς σχέδιο και χωρίς, παραλαμβάνω, να έχει προηγηθεί στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς συμφώνησε μαζί μας το Σεπτέμβριο του 2013. όπως ανακοίνωσε και η Επιτροπή Αναφορών στα μέλη της, μετά άλλαξε γνώμη. Γιατί άλλαξε γνώμη, γιατί πήρε απάντηση από την Ισπανική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα ε, εκφράστηκε η άποψη της κυβέρνησης της Εστρεμαδούρας σε αυτή την απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν άλλαξε άποψη και δέχθηκε τα νομικά επιχειρήματα της κυβέρνησης της Εστρεμαδούρα. που είναι όμως εντελώς ε, αστήρικτα, αβάσιμα. Για να σας εξηγήσω τι γίνεται. Αν υποχρεούται κάποιος να κάνει αυτή τη μελέτη ε, στρατηγικού περιβαλλοντικού αντικτύπου και προσποιείται ότι αυτό δεν χρειάζεται αφού δεν έχει φτιάξει κάποιο σχέδιο. Μα αφού δεν έχει φτιάξει σχέδιο για να μην κάνεις αυτή τη μελέτη, πρόκειται για φάρσα, πρόκειται για ανέκδοτο. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικυρώνει και να ε, επιτρέπει τέτοια πράγματα. Απαιτούνται από τη σήμανση τόσο και από την οδηγία οι μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου. Και βλέπουμε ότι δεν γίνεται ούτε σχέδιο ούτε τέτοια μελέτη και απλά υπογράφονται τα νομοσχέδια, τα διατάγματα, οργανώνεται η διαδικασία η διοικητική για να δοθεί έγκριση για την κατασκευή ενωλικού πάρκου και έτσι πηγαίνει. Αλλά ε, κάρτα πρόκειται για ένα πανδαιμόνιο, για ένα χάος. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, δεν υπάρχει καμία εκτίμηση αντικτύπου. Έτσι παραβιάζεται βέβαια η σύμβαση του όρχους από την κορυφή μέχρι μέχρι τη βάση όλοι, όλες οι διατάξεις της σύμβασης ε, και νομίζω ότι υπάρχουν και τουλάχιστον άλλες οκτώ χώρες που δεν έχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδηγία της ε, και η Επιτροπή Συμμόρφωσης της Σύμβασης του Άρχους τα καταδικάζει όλα αυτά. Επομένως, για να μην μακρηγορώ, πρόκειται για μια πραγματική καταστροφή για την Εστρεμαδούρα που έχει 80.000 ε, γερανούς, πουλιά γερανούς. Ίσως κάποιοι θα λένε ότι είναι και 120.000. Είναι ε, ένας τόπος στον οποίο χυμάζουν. Είναι μαύρη πελαργή πέντε είδη ε, αετών, ο βασιλικός αετός, ε, αυτοκρατορικός, συγγνώμη, ο χρυσός, ο χρυσαετός και άλλα είδη. Και το πουλί αυτό που πιάνει ε, τα φίδια και πάλι και άλλα είδη. Ε, γήπες, τρία είδη που το ένα είναι μάλιστα και απειλείται και με εξαφάνιση, ο Αιγυπτιακός γήπας. και άλλα ιδέα των red kites, black kites. Πρόκειται για ε, μια, τεράστια, μια περιοχή με τεράστια ποικίλια πανίδας. Και όλα αυτά απειλούνται τα είδη λόγω των αιωλικών πάρκων. Χάνονται είδη πτηνών, ε, είδη άγρας ε, πανίδας. Αν θέλουμε να βάλουμε όλα αυτά τα αιωλικά πάρκα στην Εστρεμαδούρα, θα προκαλέσουμε βιολογική καταστροφή. Και αν αυτό το κάνουμε και χωρίς στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα. Αυτά σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα. 14 είδη προστατευόμενα, απακτικά είδη. Έχουμε και κάποια ελουροειδή, οι λίγκες, οι βυρικοί λίγκες, ε, που είναι από τα πιο απειλούμενα είδη, ε, υπάρχουν στην Εστρεμαδούρα. Λοιπόν, ε, προβλήματα που υπάρχουν. Έχουμε περιχητική και χαμηλή συχνότητας χορύπανση. Όλα αυτά επηρεάζουν αν ο Λίγκα, παραδείγματο χάρη, δεν ακούει το θύραμά του, ε, γιατί κυνηγάει τη νύχτα με τα αυτιά του, αν δεν μπορεί να το ακούσει, δεν επιβιώνει. Άρα πλήρη αντίφαση εδώ. Βιολογική καταστροφή λοιπόν συντελείται, θα συντελεστεί σε αυτήν την ε, περιοχή της Τρεμαδούρας εάν εφαρμοστούν αυτά τα προγράμματα. Εμείς ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει ε, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να εφαρμοστεί αρχή της προφύλαξης και να παραλύσουν αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί ήδη από την ε, κυβέρνηση της Τρεμαδούρα και να γίνει κατεπηγόντως μάλιστα αυτό, διότι πραγματικά δεν αφορά μόνο την Εστρεμαδούρα το πρόβλημα ή την Ισπανία, αλλά και ολόκληρη τη βιοπικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν εφαρμόζουμε τον νόμο, εάν δεν απαιτούμε τη δεξαγωγή των μελετών στατικού περιβαλλοντικού αντικτύπου και την εφαρμογή των διατάξεων τη Σύμβαση του ουσιαστικά παραβιάζουμε την νομοθεσία και δίνουμε την εντύπωση ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι υπεράνω του νόμου, που δεν είναι όμω. Και δεν βοηθάμε έτσι. Γιατί μεγαλώνει το αντιευρωπαϊκό αίσθημα στην ε, Ευρώπη. Πρέπει να το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάρεκ. Α, όχι, συγγνώμη, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προεδρεύω από τις 9 η ώρα το πρωί. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον Τάνιελ Φερνάντε Κόμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον αναφέροντα για την έκθεση των γεγονότων που είναι αντικείμενο της αναφοράς αυτής όπως πολύ καλά τα είπε και ο αναφέρον, ουσιαστικά μιλάμε για παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την έγκριση και την ανάπτυξη ε, του αιωλικού σχεδίου, του σχεδίου αιωλικών πάρκων στην Εστραμαδούρα. Πρέπει να πω βέβαια, ε, σε αντίθεση με αυτά που είπε, αναφέρουν ότι εμείς λάβαμε καταγγελία ε, την διαβεβάσαμε στην Επιτροπή Αναφορών που είχε να κάνει με την ίδια εξαγωγή μελέτη στρατηγικού περιβαλλοντικού αντικτύπου για το ελληνικό σχέδιο της Εστρεμαντούρα το οποίο εγκρίθηκε με διάταγμα το 192 του 2005 συγκεκριμένα που μετά υποκαταστάθηκε από το 160 του 2010. Ε, δύο διατάγματα λοιπόν που ρύθμιζαν ε, τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών ε, ανοίγησης αιωλικών πάρκων στην Εστρεμαδούρα και έθεταν, μάλλον ανέφεραν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και διαδρόμους και ρύθμιζαν την όλη διαδικασία και το όλο σχέδιο για την δημιουργία αιωλικών πάρκων. Όπω είπε και αναφέρω, μέχρι στιγμή η Εστρεμαδούρα δεν έχει κανένα τέτοιο αιωλικό πάρκο. Αφού λάβαμε την καταγγελία λοιπόν και την αναφορά, σας τη διαβάσαμε όπω είπαμε, και ήρθαμε σε επαφή με τις ισπανικέ Αρχές. Μέσω του EU Pilot, ε, μια ηλεκτρονική εφαρμογή, ζητήσαμε λοιπόν πληροφορίες για την καταγγελία που είχαμε λάβει από τους καταγγέλλοντες και αναφέροντες. Υπήρξε μια ανταλλαγή ανακοινώσεων με στόχο εθελουσίως οι ισπανικές αρχές ε, να θέσουν τέρμα σε αυτές τις ε, ικαζόμενες παραβάσεις. Λάβαμε τις ε, πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές, λάβαμε υπόψη και τις πληροφορίες που είχαμε λάβει από τους αναφέροντες και τους καταγγέλλοντες και κάναμε την προκαταρκτική μας ανάλυση που μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πράγματι πρόκειται για ένα σχέδιο, για ένα έργο δυνάμει τη οδηγία 42-2001. Έπρεπε να γίνουν δηλαδή μελέτε στρατηγικού περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αποφασίσαμε λοιπόν να κινήσουμε διαδικασία επί και στείλαμε και την επιστολή προειδοποίηση στην Ισπανία στις 25 Απριλίου του 2013. Και εκεί καλούσαμε τις Ισπανικές Αρχές να διαβάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις παρατηρήσεις που έκριναν απαραίτητες σε σχέση με τα καταγγελόμενα και σχετικά με τις καζόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας που εμείς όπως είπα διαπιστώσαμε με την προκαταρτική μας ανάλυση ότι στέκει πράγματι υπάρχουν παραβάσεις. Στην απάντησή τους οι Ισπανικές Αρχές τουλάχιστον ε, με βάση τις υπηρεσίες της ε, Κομισιόν ε, επιβεβαιώνουν ότι αυτό το αιωλικό ε, σχέδιο δεν εμπίπτει από εφαρμογή για τι μελέτε στρατηγικού περιβαλλοντικού αντικτύπου σχέδιων και προγραμμάτων. Το άρθρο 2 τη εν λόγω οδηγία οδηγία 2042 ορίζει ποια είναι τα σχέδια, ποια είναι τα προγράμματα που υπόκεινται στη στρατηγική εκτίμηση. Και συγκεκριμένα το άρθρο 2 θεσπίζει δύο προϋποθέσεις σορευτικές, που σημαίνει ότι και οι δύο θα πρέπει να ε, εκπληρούνται, ούτως ώστε ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο να υποβληθεί σε μελέτη στρατηγικού περιβαλλοντικού αντικτύπου. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να πρόκειται για σχέδια προγράμματα που η έγκριση ή η υιοθέτησή τους ε, γίνεται από περιφερειακή εθνική τοπική αρχή και δεύτερη υποχρέωση, δεύτερη προϋπόθεση να απαιτείται από ρυθμιστικές νομικές ή διοικητικές διατάξεις. Στην προκειμένη περίπτωση, οι Ισπανικές αρχές μας ε, τεκμηρίωσαν επαρκώς ότι δεν υπήρχε κανένας ε, διοικητικός, ρυθμιστικός, νομικός κανόνας που να απαιτεί την ανάγκη εκπόνησης σχεδίου, αιωλικού σχεδίου. Ούτε σε εθνικό επίπεδο, ούτε σε περιφερειακό επίπεδο, επομένως, ε, όπως το εξήγησε και ο αναφέρον, στην Ισπανία έχουμε χιλιάδες ανεμογεννήτριες χωρίς να υπάρχει εθνικό αιωλικό σχέδιο. Και περισσότερες αυτόνομες περιφέρειες έχουν αιωλικό σχέδιο παρόλα αυτά. Η αυτόνομη περιφέρεια της Στρεμαδούρα εξήγησε ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν εγκρίνει την εγκατάσταση ολικών πάρκων στην επικράτεια της Εστραμαδούρα εφαρμόζοντας ε, την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία. Οι αρχές λοιπόν τη Αστραμαδούρα εξηγούν ότι πρόκειται για την έγκριση διαταγμάτων που συνεπάγεται απόφαση αυστηρά οικονομικής πολιτικής ε, εντός των αρμοδιοτήτων ε, τους για την νοσονομική πολιτική. Στόχος δηλαδή ήταν μέρος των κερδών από την εγκατάσταση ε, τέτοιων ε, ανεμογεννητριών θα πήγαινε ε, πίσω στην κοινωνία της Εστρεμαδούρα, που είναι αγροτική κοινωνία, δεν έχει μεγάλες βιομηχανίες η Στρεμαδούρα. Θεωρούσαν λοιπόν ότι με αυτό το σχέδιο τα κέρδη της αιωλικής ενέργειας θα μετακίνηταν στην κοινωνία. Και αυτό είναι θεμητή ε, βρίσκεται στην εκτική ευχέρεια της, ε, των αρχών της Τρεμαδούρα. Στο πείτε λοιπόν ότι πράγματι δεν είναι ένα σχέδιο που επιβάλλεται από νομοθετικές διοικητικές διαδικαστικές ε, διατάξεις. Οι Ισπανικές αρχές όπως και να έχει έδειξαν ενδιαφέρον να προχωρήσουν σε παρέκκληση σε, για αυτό το σχέδιο, επειδή έχουν αλλάξει οι συγκύρια στην Ισπανία από τότε που εγκρίθηκε αυτό το σχέδιο. Οπότε και η, ενεργεια, η αιωλική ενέργεια μεταξύ των άλλων ανανεώσιμων έπαιρναν επιδοτήσεις και μετά την χρηματοοικονομική κρίση που έπληξε με δραματικό τρόπο την Ισπανία, άλλαξε η συγκύρια αυτή. Έπαψαν να δίνονται επιδοτήσεις σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Άρα, Κατά συνέπεια αυτού υπήρξε μειωμένο ενδιαφέρον από τους εργολάβους ε, να προβούν ε, στην εγκατάσταση ολικών πέρκων στην Εστρεμαδούρα και οι αρχές της Εστρεμαδούρα ανακοίνωσαν ότι είναι διατεθειμένες ε, να το ακυρώσουν αυτό το αιωλικό σχέδιο. Έτσι και έπραξαν, ανακοίνωσαν στην Κομισιόν ότι το αιωλικό σχέδιο της Εστρεμαδούρα ακυρώνεται, αναστέλλεται μάλλον και θεωρούμε πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρήζει κλεισίματος πια η αναφορά αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Απευθύνομαι τώρα στους ε, ευρωβουλευτές. Ο Γιάρκη είναι ο πρώτος στο κατάλογό μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω την αίσθηση ότι μόλις ακούσαμε δύο ε, αντιφατικές παρεμβάσεις. Ο αναφέρον κατηγορεί τις Εθνικές ε, Τοπικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες και τώρα ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι εργασίες. Ίσως θα είναι χρήσιμο λοιπόν Ίσως θα πρέπει να φροντίσουμε αναφέρω, να λάβει το υλικό ώστε να καταλάβει τι δουλειά έχει γίνει σχετικά με αυτό το αιωλικό πάρκο. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι στο τέλος της παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσαμε ότι έχουν αλλάξει τα σχέδια, οι εξελίξεις τώρα έχουν πάρει άλλη τροπή. Δεν είμαι βέβαιος λοιπόν πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε, διότι από τη μία μου φαίνεται ότι αυτή η αναφορά δεν ισχύει πια, διότι ε, δεν ισχύει πια το αρχικό σχέδιο. Από την άλλη ακούσαμε Απ' την άλλη ακούσαμε ότι δεν έχει γίνει συγκεκριμένη ανάλυση αντικτύπου. και ότι δεν έχουν δοθεί τα στοιχεία από τις τοπικές ε, αρχές ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίλημα αντιμετωπίζω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Ε, Πρόεδρο, ε, δεν υπέροχο το ότι είμαστε όλοι άνθρωποι, ακόμα και εσύ, Γιάννη, Και είναι πράγματι πολύ δύσκολα τα θέματα αυτά. Κύριε Στέλκαμπρά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ έχω μπερδευτεί. Πολύ. Θα ήθελα, για παράδειγμα, να γνωρίζω. Το Πατρινόμονιο ε, Κουλτουράλ Διεξτρεμαδούρα είναι ιδιωτικό φορέα, είναι δημόσιο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε εάν μιλάνε στο όνομα κάποια ε, κυβέρνηση, ε, τοπικής κάποιες αρχής τοπικής ή εθνικής ή αν είναι ιδιωτικός φορέας. όχι, είναι μια ένωση ιδιωτών με στόχο να προστατεύσουμε την κληρονομιά της Εστρεμαδούρας. Επειδή είναι τόσο ε, βαρύγδουπο το όνομα, είναι περίεργο που ε, είναι όνομα ενός ε, ιδιωτικού οργανισμού, αλλά το δέχομαι αυτό, δεν έχω καμία αντίρρηση, απλά ήθελα να το γνωρίζω. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε κάτι περίεργο κατά τη γνώμη μου, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδήγησε σε αλλαγή της πολιτικής ε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό δεν ισχύει ακριβώς, διότι αυτή η αλλαγή έγινε μετά το 2012. όπου υπήρχε κρίση, αλλά όχι τόσο σοβαρή, η πραγματική κρίση χτύπησε το 2008, 2009, 2010. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση στην Ισπανία στήριζε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είδαμε λοιπόν επενδύσεις Αυτό άλλαξε επειδή προέκυψαν κάποια νομικά προβλήματα για τους επενδυτές. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ίσως μια κρυφή ατζέντα, αλλά η βασική μου ανησυχία είναι ότι δεν υπάρχει τεχνική αξιολόγηση στην ε, Εστρεμαδούρα. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνει τέτοια αξιολόγηση. Αυτό είναι τεχνικό θέμα. Γι' αυτό Προτείνω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, να λάβουμε τουλάχιστον την αξιολόγηση. Υπάρχει λοιπόν ή όχι τέτοια τεχνική αξιολόγηση. Προτείνω λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή. Ναι, και για μένα είναι πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Είναι σαν ε, να υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, αλλά ε, διαπιστώνεται ότι ο Ισπανός διαμεσολαβητής ε, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να έχει γίνει στρατηγική ε, μελέτη επιπτώσεων, κάτι που δεν έχει γίνει. Υπάρχει απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012 και το 2013, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ισπανία δεν ε, πληρεί τις υποχρεώσεις της ε, σύμφωνα με την οδηγία αυτή και συνεπώς έχει στείλει επιστολή επίσημη τον Απρίλιο του 2013 στην Ισπανία. Αλλά εκεί τελειώνουν οι πληροφορίες που έχω. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ε, αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει επικαιροποιημένες πληροφορίες όπου να αναφέρει ποια είναι η απάντηση των Ισπανικών Αρχών το 2013 και έκτοτε, διότι φαντάζομαι ότι θα συνεχίστηκε ο διάλογος αυτός για κάποιο διάστημα. Εγώ εκεί καταλήγω. Συμφωνείτε? Ωραία. Σας ευχαριστώ. Και σας ξαναδίνω το λόγο. Είσαστε ικανοποιημένος με τη λύση αυτή. Ναι, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Είχαμε μια δεύτερη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιο μακροσκελή, στην οποία συμφωνεί με τα επιχειρήματα της Ισπανικής κυβέρνησης. Και γι' αυτό έχουν μπερδευτεί πολλοί, διότι η επιχειρηματολογία της Ισπανικής κυβέρνησης που ε, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαν να προσπαθεί να παρακάμψει τα στοιχεία. Μιλάει για λεπτομέρειε, το διάταγμα που υιοθετήθηκε σύμφωνα με τον τάδε νόμο, υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει σχέδιο. Ε, νομίζω ότι προσπαθεί να θολώσει τα νερά. Και σκοπός είναι ακριβώς να μπερδέψει τον κόσμο ώστε να μην γνωρίζουν τι πρέπει να αποφασίσουν. Αλλά είναι σαφέ ότι δεν έχει υπάρξει στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση, κάτι που απαιτείται από τον νόμο, από τον κοινοτικό, αλλά κυρίως από την σύμβαση του όρκους ε, και κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Είναι λοιπόν απόλυτα ξεκάθαρη η κατάσταση. Θα πρέπει να γίνει παραδεκτή, να κρυθεί παραδεκτή αυτή η αναφορά και θα πρέπει η κυβέρνηση της Ισπανίας να πει στην τοπική κυβέρνηση της Εστρεμαδούρα ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί στρατηγική αξιολόγηση ε, ε, των επιπτώσεων, διότι προσπαθούν να θολώσουν τα νερά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις επιπλέον πληροφορίες. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που ζητάμε από την Κομισιόν είναι να βγάλει άκρη, να μας εξηγήσει τα πράγματα γραπτός, διότι γραπτός πρέπει να το δούμε. Αλλιώς ε, δημιουργείται σύγχυση όταν απλά ακούμε τις πληροφορίες και θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή ε, δύο μελών που δυστυχώς ε, δεν είναι παρόντες ε, σήμερα το απόγευμα. Γι' αυτό το θέλουμε γραπτό Έτσι θέλουμε λοιπόν όλες τις πληροφορίες επικαιροποιημένε από την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο κάτι που ανέφερε η Ορνηθολογική Επιτροπή πρόσφατα, είπε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν πλέον διότι η πολιτική έχει αλλάξει, δεν γίνονται πλέον ε, ε, επιδοτήσεις ε, για την αιωλική ενέργεια στην Ισπανία, αλλά το γεγονό είναι ότι τα νέα αιωλικά πάρκα εγκρίνονται στην Εκτρεμαδόρα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή κάτι παλιό. Δεν υπάρχει σχέδιο. Νέα αιωλικά πάρκα εγκρίνονται αυτή τη στιγμή στην Εκτρεμαδόρα χωρίς κανένα σχέδιο και χωρίς καμία εκτίμηση αντικτύπου το οποίο θα τροφοδοτήσει και τη δική μας απόφαση. Συγγνώμη κύριε Τερικαμπράς, αλλά ενισχύει ή ε, μάλλον αυτό ε, υποστηρίζει και την αποφασή μας να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ζητήσουμε ε, λεπτομερείς πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να προχωρήσουμε και μια εκτίμηση να ζητήσουμε, λίγο ο κύριος Ναι, και με αυτό θα ασχοληθούμε στην ερώτησή μας προς την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Περνάμε στο αρθρό 18 Αναφορά 1056 του 2013 του Κέβιν Κόρκεν, Ιρλανδού, που αφορά την κατασκευή ανεμογεννητριών στην κομιτεία του Κόρκ στην Ιρλανδία. Ο αναφέρον βρίσκεται εδώ, ο κύριος Κόρκεν, και σας δίνω το λόγο. Για πέντε λεπτά, όχι παραπάνω παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Γκέρα είναι ένα κομμάτι ενός αλουβιακού δάσους που βρίσκεται κοντά στο Κόρκ στη Δυτική Ιρλανδία. Είναι ε, μια από τι σπάνιε περιοχές ε, εύκρατου ε, δάσους των βροχών και επιστημονικά είναι ένα αλουβιακό δάσος που δημιουργήθηκε μετά από την εποχή των Παγετώνων και είναι από τα σπάνια ανάγκη δάση που έχουν παραμείνει ε, τέτοια τροπικά δάση στην ε, Δυτική Ευρώπη ε, και βρίσκεται υπό προστασία δυνάμει της οδηγίας 92-43 της ΕΟΚ. Η μοναδική δασόδης περιοχή στη συμβολή των ποταμών Λί και Τούν όπου σχηματίζεται ένα εσωτερικό δέλτα δασοδών νησών μεταξύ ενός λαβυρίνθου ε, διακλαδώσεων ε, ρευμάτων. Τα νησιά αποτελούνται από προσχωσιγέννη ύλη ε, και συγκρατούνται ακέραια από τις ρίζες των δέντρων, οπότε η επιβίωση εξαρτάται από την η χρηστή διαχείριση των υδάτων στην λεκάνη απορροής. Τα τελευταία χρόνια η υδρολογία του ποταμού Τόν ε, έχει υποβαθμιστεί σημαντικά λόγω της συνεχούς καταστροφής των οικολογικών παραμέτρων του ποταμού ε, πιο ψηλά από το δάσος. Αυτές ε, οι αφύσικες πλημμύρες έχουν δημιουργήσει ε, κατάρρευση του οικολογικού συστήματος. Ε, βλέπουμε πάρα πολλά δέντρα που πέφτουν και νησιά που συνδείχεται είναι κάτι ορατό και τα κανάλια ε, αποξηραίνονται ενώ τα ρεύματα μαζεύουν υλή. Μία εταιρεία αιωλικών πάρκων έχει ένα έργο να αναπτύξει ένα αιωλικό πάρκο στο την περιοχή αυτή. Αλλά επειδή το έργο έχει χωριστεί μεταξύ πολλών μικρών εταιρεών, ε, αξιολογείται το έργο ε, και όχι σωρευτικά. Οπότε θεωρείται ότι δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις. Τα αιωλικά πάρκα αυτά ε, πρόκειται να εγκατασταθούν σε ανέγγιχτες περιοχές εδώ και εκατοντάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια ε, και τα οικοσυστήματα αυτά λειτουργούν ως τεράστιοι σπόγγοι που απορροφούν το βρόχινο νερό. Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις με αμφισβητήσιμους τεχνητούς μηχανισμούς που έχουν αποτύχει επανειλημμένως σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αλλά ε, φαίνεται ότι αυτές οι, αυτοί οι ισχυρισμοί ικανοποιούν τις απαιτήσει ε, ε, της οδηγίας για τα οικοσυστήματα, για τα ενδιατήματα. Έχει παρατηρηθεί ήδη τι τρομακτικές που είναι οι επιπτώσεις ε, ε, στα οικοσυστήματα από τέτοια αιωλικά πάρκα. πάρκα θα δημιουργηθούν πλημμύρες στην προκειμένη περίπτωση και θα επιτείνουν τη διάβρωση του Δέλτα του Γκέραχ. θα πρέπει να κάνουμε για να προστατευτεί το δάσος, αλλά όλα μας οι εκκλήσεις έχουν ε, παραβλεφθεί ε, πλήρως. Και στην περίπτωση αυτή η οδηγία για τα διατήματα δεν εφαρμόζεται επαρκώς. Τώρα, με αυτή την αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η πρώτη φορά που τίθεται αυτό το θέμα εδώ, αλλά ουσιαστικά θα προεκτέ απλά για μια άσκηση ε, δημοσίων σχέσεων στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναφορών. Συμπερασματικά λοιπόν δεν γίνεται καμία προσπάθεια πρόληψης της ε, καταστροφής ε, του δάσους που είναι παραβίαση του άρθρου 62. Δεν υπάρχουν ορθές πρακτικές διαχείρισης στις λεκάνες απορροής και αυτό αποτελεί παραβίαση του άρθρου 6.3. Οπότε κάνω έκκληση στην Επιτροπή Αναφορών να εξετάσει προσεκτικά τη σοβαρότητα της αναφοράς μου, διότι ο σκοπός δεν είναι απλά να προστατευτεί η γκέρα, αλλά η αικαιρεότητα των ενδιατημάτων και της εφαρμογής της οδηγίας για τα ενδιατημάτα στη δική μου χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τζουράστη, όχι, πάλι το ίδιο κάνω. Η, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κύριος Μάικλ Ομπράιεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και να ευχαριστώ και τον κύριο Κόρκορεν για την ε, παρουσίασή του ε, έτσι όπως παρουσίασε τα ζητήματα. Ζητώ συγγνώμη γιατί ο συνάδελφος μου, η συνάδελφος μου Λόγκ που ασχολείται με αυτό το φάκελο έχει τραυματιστεί και δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ σήμερα. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η περιοχή για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη έχει συμπεριληφθεί στην οδηγία για τα ενδιατήματα. Η περιοχή αυτή έχει υποστεί τεράστια ζημιά ήδη στο παρελθόν. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι που έγινε δεκαετία του 50 λόγω ενός μεγάλου ε, υδροελεκτρικού έδρου που πλημμύρισε και καταστρέψε πάρα πολλές περιοχές. Εξακολουθεί όμως να έχει πολύ ψηλή αξία διατήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο ε, διαχείρισης, ε, αποκατάστασης και προστασίας. Ε, όταν πρώτο αναφέρθηκε, πρώτο υποβλήθηκε αυτή η αναφορά, ο αναφέρον είχε γράψει και στην Κομισιόν και εμείς το, πήραμε το θέμα αυτό πολύ στα σοβαρά ε, και το συζητήσαμε με τις Ιρλανδικές Αρχές. Είχαμε μια αναφορά το 2014 η οποία εξέταζε τα επί της ουσίας ζητήματα όσον αφορά την προστασία και τη διαχείριση και σε σχέση με το ρόλο των τοπικών αρχών του αναπτυξιακού σχεδίου της Κομιτείας αλλά και σε σχέση με οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία είχαμε όσον αφορά την ανάπτυξη της αιωλικής ενέργειας. Και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Φυσικά το ζήτημα της διαχείρισης ε, είναι κεντρικό για την προστασία αυτού του τόπου και ε, συνεχίζονται ακόμη οι συζητήσεις ε, με τις ελληνικές αρχές και ελπίζω ο κ. Κόρκαν να αναγνωρίσει ότι κάτι κινείται για τη δημιουργία ενός σχεδίου διαχείρισης το οποίο θα αντιμετωπίσει τα υδρολογικά ζητήματα τα σημαντικά υδρολογικά ζητήματα και φυσικά πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα διότι υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων, των πλημμυρών, αφορούν και άλλα νομοθετήματα. Οπότε οι εργασίες αυτές ε, βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτό είναι θετικό αποτέλεσμα σε σχέση με την αναφορά και με τις έρευνες της ε, Κομισιόν. Οι Ιρλανδικές αρχές ε, επιβεβαίωσαν ότι το αναπτυξιακό σχέδιο της Κομιτείας πράγματι λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσει τις οδηγίες για τα ενδιατήματα σε σχέση με την ανάγκη μεταξύ άλλων επαρκούς αξιολόγησης. Το ζήτημα της ανάπτυξης ανάντιν και το ζήτημα της ανάπτυξης ελικών πάρκων και εγκατάστασης ελικών πάρκων υποκείται στην διαρκή ε, διαδικασία σχεδιασμού στην Ιρλανδία. Τώρα το κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος για μια περιοχή του Natura 2000, αυτό πρέπει να, εκεί πρέπει να γίνει η απαρχής αξιολόγηση, να εξεταστεί ο κίνδυνο και να αποτιμηθεί. Αυτό έχει γίνει και περιλαμβάνει και έναν ε, ειδικό υδρολόγο, αλλά λαμβάνει υπόψη τα σχόλια του κ. Κορκάνη σήμερα όσον αφορά το ζήτημα των μικρών εγκαταστάσεων που η καθεμία δεν αποτελεί κίνδυνο αλλά οι οποίε ορευτικά όμω αποτελούν κίνδυνο οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το κοιτάξουμε να το εξετάσουμε περαιτέρω το ζήτημα δεν έχει κλείσει και θα υπάρξει κάποια έκκληση ξανά στο ελληνικό σύστημα. Πιστεύω ότι τηρούνται οι απαραίτητες διαδικασίες και φυσικά όσο ε, ε, υπάρχει αυτή η διαδικασία που τρέχει δεν θέλουμε να παρεύουμε άλλο. Μπορεί να ζητήσουμε περαιτέρω εξηγήσει. Θα θέλαμε όμως αν υπάρχουν άλλα νέα ζητήματα, ή ζητήματα που δεν έχουμε καλύψει και εκεί υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για μη συμμόρφωση, εκεί ευχαριστώ να ε, θέσουμε ξανά το θέμα στι Ιρλανδικέ αρχέ. Ε, πιο γενικά, ήθελα να πω ότι συνεχίζεται η συζήτηση με τι Ιρλανδικέ ε, αρχέ για το θέμα του καθορισμού και της ε, εφαρμογής των μέτρων διατήρησης γενικότερα. Έχουμε μια διαδικασία δηλαδή που τρέχει, έχουμε πάρει πολύ σοβαρά το θέμα αυτό και φυσικά οποιοδήποτε θέμα εκκρέμει ή προκύψει, ευχαριστώ να το ερευνήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ. Thank you Εμείς σας ευχαριστούμε. Τώρα, τέλος. Και συγγνώμη που κάθεστε. Κύριε Γιουράστη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να αναφέρω τη στήριξη της GUNGL στην ε, αναφορά Κόρκοραν και αυτό ρητός εξ ονόματος ε, συναδέλφου Λιέτ που είναι από το Συνφέν δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε. Θεωρούμε ότι είναι σωστό ένα προρθένο τροπικό δάσος, αλουβιακό δάσος πρέπει να διατηρηθεί, να προστατευτεί, το είπε ο αναφέρον, το λέει και η Κομισιόν ότι είναι μοναδικό μέρος αυτό ε, στην Ευρώπη. Δυστυχώς σήμερα απειλείται, παρότι πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή, δυνάμει της οδηγίας για τα ενδιατήματα, για τους οικοτόπους και Φαίνεται ότι δεν εφαρμόζονται σωστά εδώ οι διατάξει οδηγία. Μα εξήγησε ο κύριο Κόκοραν πώ απειλείται το μέρο αυτό. Η Γκουεντζέλ ακριβώ γι' αυτό θα ήθελε να ζητήσει από την Επιτροπή Αναφορών να αφήσει ανοιχτή την αναφορά. Θα ήθελα επίση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει ιδίω τα εδάφια 2 και 3 του άρθρου 6 τη οδηγία για του Οικοτόπους που μιλάει για τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν για να διατηρηθούν οι φυσικέ ε, προστατευόμενε περιοχέ. Και θεωρώ επίση σκόπιμο η Επιτροπή μα. να αποστείλει στην Επιτροπή ΕΝΒΗ προ εξέταση το θέμα αυτό. Είμαι μέλο και τη Επιτροπή ΕΝΒΗ προσωπικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει νομίζω κατά κάποιον τρόπο ότι ακόμη απομένει δουλειά να γίνει. Χρειάζεται να συλλεγούν ακόμη πληροφορίε, ε, να γίνουν έρευνε. Γι' αυτό ζητούμε να παραμείνει ανοιχτό το θέμα. Θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, είναι ένα δάσο ιδιαίτερο και όσοι και αν, όσο και αν μικρή να είναι η αμφιβολία μας, παρόλα, ακριβώς όσο παραμένει στο και ένα ψήγμα, αμφιβολία θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό το θέμα. Ευχαριστώ. Γιάρικ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ναι, είναι σαφέ ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Αυτά που μα είπε η Κομισιόν είναι ενθαρρυντικά, σίγουρα. Από ό,τι φαίνεται κάποια πρόοδο σημειώνεται. Όμω, είναι προφανέ ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τι διάφορε περιοχέ. Είναι κάτι που είναι απαραίτητο, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και μέχρι ότου ολοκληρωθεί πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση και να μην είναι ανοιχτή αναφορά. Η ε, πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριο σε ευχαριστώ πολύ. Μετά από όλες τις παρεμβάσεις γνωρίζουμε, ή εγώ τουλάχιστον, δύο πράγματα. Πρώτον έγινε πρόοδος, η συζήτηση συνεχίζεται και βέβαια υπάρχει ανάγκη ε, της σωστής εκτίμησης και αξιολόγησης. Αν αυτά τα δύο τα προσθέσουμε, τι σημαίνει ένα και ένα κάνουν δύο, παραμένει η ανάγκη να μην ανοιχτή η αναφορά. Είναι σαφές. Ευχαριστώ. Η Ελεονόρα τι έχει να μας πει. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά διότι επίσης μου φαίνεται ότι διακρίνω μια κατάσταση ή μάλλον μια από τις στρατηγικές που συχνά εφαρμόζονται για τα μεγάλα έργα. Δηλαδή τα κατακαιμαρτίζουν σε μικρά κομματάκια ώστε να περάσουν πιο εύκολα από τη φάση έγκρισης. Είναι μια τυπική λοιπόν περίπτωση, οπότε πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά αυτή και να την εξολογήσουμε να την αποτιμήσουμε, διότι στρατηγικές τέτοιου τύπου δεν είναι παραδεκτές ε, ειδικότερα σε συνθήκες περιβαλλοντικές αυτού του τύπου που πρέπει να προστατεύσουμε. Now. Μάλιστα. Κύριε Κόρκονεν. γρήγορα παρακαλώ. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω τα σχόλια για τα σχόλια υποστήριξη. Και εγώ προσπαθώ ε, να πετύχω κάποια πρόοδο μεμονωμένα. Λίγο πριν φύγω από την Ιρλανδία με το αεροπλάνο είδα ε, τα μηχανήματα στο φυγή του ποταμού ουσιαστικά, ε, είδα φορτηγά, ε, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται ακριβώς, είναι εκ υπάρχουν γραφειοκρατικοί λόγοι, φοβούμε πάντως. Μην κλείσει η αναφορά και ξανά εγώ μετά σε δύο χρόνια εδώ να λέω τα ίδια και να εκλυπαρώ για μια ακόμη φορά για τη βοήθειά σας, για την προστασία αυτού του κοσμήματος. Ο κ. Στερικάμπρας. κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, ποιος είναι ποιος, με ενδιαφέρει πάντα. Εσείς τι είστε, είστε ιδιώτης που προασπίζεστε από μόνο σας. Δεν σας στηρίζει κανείς, δεν έχετε καμία υποστήριξη. Με είναι εξαιρετικό αυτό. Ή έχετε κάποια υποστήριξη. Κύριε Σκόρκορα, όχι, να σας εξηγήσω. Αυτό το δάσος πριν το καταστρέψει αυτό το ρεκτικό φράγμα, καλύπτει αρκετά χιλιάδες εκτάρια. Η οικογένειά μου, η οικογένεια της μητέρας μου και άλλοι ε, ζούσαμε εκεί, στα δάση αυτά και μας ανάγκασαν να φύγουμε. Μας μετεγκατέστησαν αλλού. Και εγώ ενημερώθηκα από τη μητέρα μου, από τους παππούδες μου για το δάσος Πήγα στο σχολείο και μελέτησα και τη θα δάση και τα τελευταία 25 χρόνια αγωνίζομαι για την προστασία αυτού του δάσους και με τιμά ιδιαίτερα από το γεγονός ότι μπορώ εδώ να σας μίσω σε ο τελευταίος των Μοϊκανών. Σας παρακαλώ να σώσετε ε, αυτό το προγονικό δάσος και να προστατεύσετε και την ακαιρεότητα της οδηγίας για τα ενδιατήματα για τα οικοσυστήματα για να μπορώ να φύγω από εδώ λέγοντα ζήτω η δημοκρατία, ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you very much. And this is... Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο τέλειος ο τρόπος να κλείσουμε την αναφορά. Ε, να κλείσουμε τη συζήτηση για την αναφορά αυτή, να συμφωνούμε όλοι, να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή και να ε, καλέσουμε την Επιτροπή να συνεχίσει το διάλογο με τις Ιρλανδικές Αρχές και να επανέλθουν στην Επιτροπή μας ε, με πλήρη αξιολόγηση. Θα ήθελα πάρα πολύ να θέσω προθεσμία. Μπορεί το 12 να ακούγεται τρελό, αλλά πριν το καλοκαίρι ίσως, μήπως κατά τη διάρκεια της Άνοιξης να έχουμε μια προθεσμία για να έχετε το χρόνο που χρειάζεστε. Δεν θέλω να σας πιέσω, αλλά παρακαλώ μην περιμένετε υπερβολικά πολύ. Και θα θέλαμε πολύ, αν είναι δυνατόν, να λάβουμε γραπτό στην απάντησή σας. Και είμαι βέβαιη ότι είναι δυνατόν να τη λάβουμε γραπτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία τώρα που θα επιστρέψετε στην Ιρλανδία. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια συμβουλή για ένα ε, βιβλίο που λέγεται «Ο άντρας που φύτευε δέντρα» που ε, έγραψε τη δεκαετία του 50 ένας εξαιρετικός Γάλλος συγγραφέας και μου θυμίζεται ακριβώς αυτόν τον άνθρωπο. Επιστρέψτε λοιπόν στο δάσος σας ε, με τις καλύτερες ευχές μας. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έτσι ολοκληρώσαμε τις σημερινές μας εργασίες. Κάποιοι από εσά επέμειναν, μείνανε εδώ. Πάλι και εγώ νομίζω ότι είμαστε εδώ από τις 9 το πρωί. Και θα τα ξαναπούμε τον Οκτώβριο, σε ένα μήνα, στις 10 Οκτωβρίου. Συνεχίστε λοιπόν ε, την ε, καλή δουλειά σας ε, και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα στο Στρασβούργο.